Καλημέρα σας. Ξεκινούμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Αναφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ε, συνεδρίασης των συντονιστών που έγινε χθες το βράδυ. Οι συντονιστές σημειώνουν ότι η μερίσια διάταξη 27 26 ε, ε, Οκτωβρίου είχε γίνει δεκτή με τη γραπτή διαδικασία και δέχτηκαν τα αιτήματα των πολιτικών ομάδων για, την, ε, για τον Ιανουάριο. Σε ό,τι αφορά την ε, ηλιακή ενέργεια και την σχετική οδηγία, συμφώνησαν να υιοθετηθεί σύντομο ψήφισμα και να υπάρξει και γνωμοδότηση για την επόμενη νομοθετική πρόταση, όπως πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συντάσεις έγιναν δεκτές με τη μορφή που τις πρότεινε η Πρόεδρος στις συμβιβαστικέ προτάσεις βέβαια. Για το Β τμήμα έχει κλείσει τον αναφορών η ατζέντα του Σεπτεμβρίου και θα παρουσιαστούν γραπτώς τα αιτήματα για να μπουν αναφορές στο τμήμα Β. Σε ό,τι αφορά τις ακροάσεις για το πρώτο εξάμεινο του 2005, λέει ο Μιλήτριο, οι συντονιστές αποφάσισαν αποστολή στη Σουηδία το Φεβρουάριο και στην Ισπανία τον Μάιο του 2017. Και θα υπάρξει νέα πρόταση για την αποστολή στο Τάραντο, που ε, λόγω έλλειψης απαρτίας δεν είχε γίνει δεκτή πριν από μια εβδομάδα. Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα του Brexit και συμφωνήθηκε την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών να συζητηθεί ξανά και να υπάρξουν ενημεριωτικά σημειώματα για το θέμα αυτό από τα αρμόδια τμήματα. Ω προ τα ερευνητικά προγράμματα για το 2017, οι συντονιστέ σημειώνουν την πρόταση που παρουσίασε το Τμήμα Πολιτικής και ορίζεται προθεσμία για την υποβολή προτάσεων μέχρι τη 17η Νοεμβρίου. Ε, σύμφωνα με την Ελεονόρα, η ομάδα εργασίας θα ασχοληθεί με θέματα παιδικής εργασίας και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα πριν από το Μάρτιο του 2017. Και θα υπάρξει συνάντηση σε διακοινοβουλευτικό επίπεδο για αυτά τα θέματα, αλλά θα αποφασιστεί στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Στηρίξαμε την οργάνωση Τη διάσκεψης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με αναπηρίες για το 2017. Αυτό το ζήτησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις αναπηρίες και ζητήθηκε η Επιτροπή Αναφορών να ε, προσφέρει στήριξη σε αυτό το γεγονός και θέλουμε να υπάρξει και μια πλατφόρμα για την ισότητα των φύλων. και ο Πίτερ θα είναι ο σύνδεσμος με αυτή την Επιτροπή των Γυναικών. Αυτά για τους συντονιστές. Περνάμε τώρα Μου λένε ότι έχει έρθει μια ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Κέντ στις Βρυξέλλες. Τους καλωσορίζουμε. Πρέπει να κάνουν μια προσωμείωση της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της ερευνητικής τους εργασίας στην τάξη. Καλώς ήλθατε. Ερχόμαστε τώρα στο, ε, στους αναφέροντες έχουμε την αναφορά για τον εξυγχρονισμό των γραμμών του τραμ στη Σλοβακία, στο Λιτόψκι. Ο αναφέρον θέλει να παραμείνει ανώνυμος. Να δώσουμε το λόγο στη Ρίτα. Στο Ρίτσαρτ Σούλικ μάλλον. Εξ ονόματος του αναφέροντος, ο οποίος και θα διαβάσει την ε, αναφορά του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι η Επιτροπή Αναφορών θέλησε πραγματικά να ασχοληθεί αυτό το, με αυτό το ζήτημα. Το 2015 υπήρξε μια αναφορά που εστάλει στην πόλη στο Δημοτικό ε, Συμβούλιο του Λιπτόφσκι Μικούλας με υπογραφή 500 ατόμων κατά της κατασκευής μιας νέας γέφυρας για την οδική κυκλοφορία και ο Δήμος αγνόησε αυτή την αναφορά και γι' αυτό οι πολίτες στρέφονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη Σλοβακία υπάρχει ένα project εξυγχρονισμού στο βορρά για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή και το στηρίζουμε ολόψυχα ολόθερμα το project της αναβάθμισης των ε, σιδηροδρομικών γραμμών. Αυτό θα ωφελήσει τους πολίτες. Όμως, όπως έχει ήδη συμβεί και στο παρελθόν, και το έχουμε βιώσει, έχουμε αυτή την εμπειρία, η πόλη, ο Δήμος επιβάλλει προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα, διότι θεωρεί ότι το, την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου ότι είναι μια ευκαιρία να χτίσει κάτι τζάμπα, δωρεάν. Και γι' αυτό βάζει οικονομικά προεπαιτούμενα. Να σας εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται. Στο χάρτη βλέπετε το τμήμα της πόλης, Λιπτόφσκι Μίκουλας, που είναι κοντά σε ένα βουνό, σε μια οροσυρά, στο βόρειο τμήμα της Σλοβακίας και χωρίζεται από το ποτάμι στα δύο. Έχουμε το βόρειο μέρος της πόλης πάνω από το ποτάμι και εκεί βρίσκονται όλες οι υποδομές της πόλης, ενώ στο νότιο μέλος από την άλλη πλευρά του ποταμιού είναι ένα σούπερ μάρκετ και ο καταβλισμός των πληθυσμών Ρωμά. Θα γίνει με την κατάσταση του πληθυσμού αυτού σε ένα άλλο μέρος της πόλης. Τι γίνεται λοιπόν με το σιδηρόδρομο. Οι σιδηρόδρομοι θα μεταφερθούν προς τον νότο και για να συνδεθεί η σιδηροδρομική υποδομή με την πόλη, ο Δήμος σχεδιάζει να χτίσει αυτή τη γέφυρα. Θα μεταφερθούν σε αυτό το ορθογώνιο που βλέπετε εκεί. Έχουμε γέφυρα με τις πράσινες γραμμές και την ενιαία και αυτή με τις τελίτσες. Υπάρχουν αυτές οι δύο γέφυρες και καλύπτουν πλήρως τις κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης όλα αυτά, ο Δήμος σχεδιάζει να χτίσει μια καινούρια γέφυρα, την κόκκινη, με τις κόκκινες βούλες που δεν υπάρχει ακόμα, ανάμεσα στις δύο υφιστάμενες γέφυρες που φαίνονται στο χάρτη με πράσινο. Οι ανησυχίες είναι πολύ μεγάλες, διότι θεωρούν οι κάτοικοι που ε, ζουν εκεί ότι η ποιότητα ζωής τους θα υποβαθμιστεί ιδιαίτερως από αυτό το project, από αυτό το σχέδιο. Οι αμφιβολίες είναι απολύτως βάσιμες και ξέρετε, αν το κοιτάξει κανείς καλύτερα, βλέπει ότι αυτή η γέφυρα δεν σχετίζεται με την νέα σιδηροδρομική υποδομή. Είναι απλά κάτι που θέλει ο Δήμος να χτίσει. Τελικά θα μειωθεί, θα υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής, γιατί υπάρχει ποδηλατόδρομος, ο οποίος φτιάχτηκε το 2014 αυτό είναι ένα διασυνοριακό project ε, στα πολλοσλοβακικά σύνορα και θα πρέπει βασικά να καταργηθεί και να καταστραφεί ο ποδηλατόδρομος προκειμένου να υπάρξει αυτή η γέφυρα. Θεωρούμε ότι οι φήμες που κυκλοφορούν είναι απολύτως βάσιμες. Η Επιτροπή Αναφορών εξέδωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο αναφέρον θεωρεί ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα εμπλακούν στην κατασκευή βεβαίως αυτής της γέφυρας και αυτό ε, τελικά είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η ιστορία και μπορεί να υπάρξει ε, ε, κακή χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων ενδεχομένω. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει γίνει αξιολόγηση αντικτύπου σε περιβαλλοντικό επίπεδο, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι δικαίωμα του κοινού να λάβει ε, πληροφορίες ε, πλήρης και σε έφθετο χρόνο για αυτό το σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση θα αναβαθμιστεί η αξία της περιοχής εκεί με την κατασκευή αυτής της γέφυρας και θα αυξηθούν και τα επίπεδα του θορύβου κατά 10 δεσιμπέλ σε μια ζώνη που είναι εξαιρετικά οικιστική και έχει πάρα πολλούς κατοίκους. είναι δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν προστασία από το θόρυβο, από τη σκόνη, από τις εκπομπές ε, λόγω της ευεβαρημένης ε, κυκλοφορίας. Θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έργα ηχομόνωσης προστασίας είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία να περιλάβει και το θέμα του θορύβου και να προταθούν και μέτρα για τη μείωση των επιπέδων θορύβου. Σε κάθε περίπτωση η γέφυρα αυτή είναι μια επένδυση φυτευτή θα έλεγα και η απόφαση για την απόφαση αρμοδιότητα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμβούλιο και συνήθως τα δηματικά συμβούλια ε, για να ε, ε, για να δεχθούν μεγάλα επενδυτικά project όπως είναι η μεταφορά των συντηροδρομικών υποδομών έχουν θέσει ως προαπαιτούμενο τα, τα, τα αντισταθμιστικά ωφέλη από την κατασκευή αυτής της γέφυρας. Γι' αυτό και θα ήθελα να κάνω την εξής πρόταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να παρακολουθεί τον κανονισμό, την νομοθεσία που διέπει ε, τις αναβαθμίσεις του δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών. Δεύτερον, την ε, υπόθεση αυτή να την εξετάσει και η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφέρει γνωμοδότηση για το κατά πόσο Μπορεί να υπάρχουν πολλές τέτοιες ε, περιπτώσεις όπου τα δημοτικά συμβούλια για να εγκρίνουν επενδυτικά project απαιτούν κατασκευή άλλων ε, ε, υποδομών και θα ήθελα και η Επιτροπή Περιβάλλοντος να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και το τέταρτο που θα ήθελα να προτείνω είναι το εξής. Άπαξ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παράσχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει επιστολή στο Σλοβακικό Υπουργείο Μεταφορών εκφράζοντας ανησυχίες για την καθυστέρηση του, της υλοποίησης του έργου των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ε, το έργο των σιδηροδρομικών μεταφορών έχει καθυστερήσει λόγω αυτής, ε, αυτού του προαπαιτούμενου που θέτει το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να το εγκρίνει και προαπαιτούμενο με το οποίο η ευρύτερη κοινότητα των κατοίκων δεν συμφωνεί και ελπίζουμε να, τελικά να μην αξιοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια για να πετύχουν σκοπούς που είναι αντίθετοι ε, ε, με, τον αρχικό προορισμό των χρημάτων αυτών. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η γέφυρα αυτή πλήττει το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χάρος Λάπιστρακ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα γιατί το να ε, τονίζουμε τέτοια ζητήματα μας βοηθά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθούμε στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στον τομέα των μεταφορών και να βελτιώσουμε την ποιότητα των σχεδίων έτσι ώστε να υπάρχει σωστή σχέση κόστους οφέλιας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που εφήγει αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, μπορούμε να πούμε ότι ήδη έχουμε θίξει αυτό το θέμα με τις σλοβακικές αρχές πολλές φορές και σε πολλές συναντήσεις και θα το κάνουμε και στο μέλλον. Όπως γνωρίζετε, η προετοιμασία αυτού του σχεδίου υποδομής είναι ένα μακροχρόνιο ζήτημα και αυτή τη στιγμή καλέσαμε τις σλοβακικές αρχές να μας δώσουν τις σχετικές πληροφορίες καθώς και αιτιολόγηση για αυτή τη γέφυρα και την κατασκευή της που αναφέρεται στην αναφορά. Όταν θα έχουμε όλες τις πληροφορίες θα τις εξετάσουμε και θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο στο θέμα σε σχέση με τη γέφυρα αυτή. Εάν οι σλοβαϊκές αρχές δεν μπορέσουν να αιτιολογήσουν την κατασκευή αυτής της γέφυρας σε σχέση με τη δημιουργία νέας σιδηροδρομικής γραμμής, τότε δεν θα χρηματοδοτηθεί αυτή η γέφυρα από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτά εντάχει από τη δική μας πλευρά και θα παρακολουθήσουμε το ζήτημα αυτό εκ του σύνεγγης για τη διασφάλιση μιας σωστής συνέχειας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα οι βουλευτές έχουν το λόγο. Ο κύριος Βαλέσα. Είπατε ότι ο Δήμος και η πόλη θέλουν να κατασκευάσουν αυτή τη γέφυρα δωρεάν και μιλήσατε για κατάφχρηση κοινοτικού χρήματος και κάπως με μπερδέψατε. Μιλήσατε επίσης και για τη μελέτη αντικτύπου και το θέμα της συγχωρήπανσης. Αυτό θα μπορούσε να απασχολήσει την Επιτροπή, γιατί πρόκειται για μία μακροχρόνια επένδυση και γι' αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε, να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Έχουμε μία περίπτωση η οποία εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Και το λέω αυτό μια και έχουμε τους φοιτητές μας οι οποίοι παρακολουθούν αυτή τη συνεδρίαση και καλό θα είναι να επισημάνουμε ότι πράγματι αυτή η υπόθεση εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ε, αναφέροντες ή την αναφέρουσα ε, για το θέμα το οποίο έχει θέσει. Ορθώς, σύμφωνα με τον κανονισμό, επιτρέπεται κάποιος αναφέρον να μην αναεξηγήσει και να μην πει το όνομά του, διότι είναι καθαρά δικαίωμά του. Και φυσικά στην περίπτωση αυτή μπορεί κάποιος βουλευτής να τον εκπροσωπήσει και ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον κύριο Σούλικ που ανέπτυξε την αναφορά. Το τρίτο θέμα είναι ότι θεωρούμε ότι η θέση της Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για μια πραγματική εξέταση της υπόθεσης, διότι είπε η Επιτροπή ότι θα παρακολουθήσει από κοντά την υπόθεση, θα την αναλύσει, θα δει εάν υπάρχουν επιπτώσεις και παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα είναι διατεθειμένη να μην χρηματοδοτήσει το project. Αυτό λοιπόν δείχνει την αποφασιστικότητα με την οποία μπορεί να δράσει η Επιτροπή μετά από ένα αίτημα ενός πολίτη. Και είναι ο σημαντικός ρόλος του δικαιώματος αναφοράς που υπάρχει και η δουλειά η οποία γίνεται σε αυτή την Επιτροπή. Το τέταρτο θέμα είναι ότι αναπτύχθηκε από τον συνάδελφο πάρα πολύ αναλυτικά και είδαμε και το διάγραμμα τις επιπτώ... οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν με αφορμή ε, την, ε, το project αυτό και τις παραβιάσεις που θα έχουμε στο πεδίο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν,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 Ε, έλεγα λοιπόν ότι ε, είναι σημαντικό το πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Επομένως η πρόταση που διαμορφώνουμε εμείς ως CCR είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να είμαστε σε επαφή με τον αναφέροντα και κυρίως με τον ε, Ευρωβουλευτή μας τον κύριο Σούλικ, να αναμείνουμε τα αποτελέσματα της ε, έρευνας που θα κάνει η Κομισιόν και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή την υπόθεση. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε στη βάση αυτή να προχωρήσουμε ε, διατηρώντας ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή. Ευχαριστώ. Ε, Θα κάνουμε την εξής πρόταση. Α, όχι, θα δώσω το λόγο καταρχήν στον αναφέροντα, στον εκπρόσωπό του για δύο λεπτά, για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που εξέφρασαν την άποψή τους για αυτή την αναφορά και την υποστήριξαν. Θα ήθελα να σας εξηγήσω τι εννοούσα για, ως προς τη ε, δωρεάν κατασκευή. Μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες είναι απαλήτως αναγκαίες για τον απότερο στόχο, δηλαδή τον εξυγχρονισμό αυτής της σιδηροτροχιάς, αυτής της γραμμής. Οι άνθρωποι όμως, οι πολίτες θα ήθελαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει το κόστος της γέφυρας που δεν εκπροσωπεί μέρος αυτού του έργου. Εγώ ήμουνα σε επαφή για ένα χρόνο με τους αναφέροντες και είδα επιτοπίως την κατάσταση και γι' αυτό τους εκπροσωπώ γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή η γέφυρα δεν είναι αναγκαία και θα μειώσει την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Πρόκειται για μία πόλη 25.000 κατοίκων. Εάν 1.600 υπέγραψαν, κάτι σημαίνει αυτό. Θα κάνουμε την εξής ε, πρόταση. Θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά όπως ζήτησαν όλοι μέχρι ότου ε, λάβετε μία απάντηση από τις σλοβακικές αρχές, αναφέρομαι στην Κομισιόν, σε σχέση με τη χρήση των ε, διαρθρωτικών πόρων και θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να μας μιλήσει για την περίοδο προγραμματισμού 14-20 για να δούμε πού εντάσσεται αυτό το σχέδιο. Θα ζητηθεί και γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Περιβάλλοντος και θα αναμείνουμε και τις απαντήσεις στην απάντηση των Σλοβακικών Αρχών. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην επόμενη που είναι η 35 κάθετος 2015 του Ανδρέα Τσόρι σε σχέση με την ε, περιβαλλοντική προστασία της ε, θαλάσσιας περιοχής σου Παλώσου στη Σαρδινία. Το λόγο έχει ο... Όχι, ο αναφέρον δεν παρίσταται. Άρα δίνουμε το λόγο στη Μαγδαλένα Προύνα, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επίτροπης. Καλημέρα σας. Από τις πληροφορίες που λάβαμε από τον αναφέροντα δεν είναι σαφές κατά ποιο τρόπο η τροποποίηση του σχεδίου διαχείρισης του Natura 2000 σε ό,τι αφορά την ε, μεταφορά της ε, εγκατάστασης μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι Ιταλικές αρχές ε, έκαναν μια, μια μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου σε ό,τι αφορά τη μετατροπή αυτή και ελήφθη η απόφαση να μην ακολουθήσει μια πλήρη διαδικασία γιατί δεν υπήρχε σημαντικός περιβαλλοντικό αντίκτυπος κατά πάσα πιθανότητα. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ε, αναφορά του αναφέροντα δεν μπόρεσε να βρει τεκμήρια για ενδεχόμενη παράληψη, ε, αγνόηση ενδεχόμενων κινδύνων για την δημοσία υγεία. Και θα θέλαμε να ενημερώσουμε και τον αναφέροντα και τους εξέτοιμους βουλευτές ότι η σχετική νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση δημοσίευσης των σχεδίων για τις εγκαταστάσεις αυτές πριν τη δημοσίευσή τους, πριν την εφαρμογή τους. Ωστόσο, δεν προδιαγράφεται το πώς θα γίνεται η διαβούλευση, ούτε προβλέπεται μια άμεση πρόσκληση του κοινού στη διαδικασία και σύμφωνα με το άρθρο 17 της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Χάρτας και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία προβλέπονται στο άρθρο αυτό και εξαιρέσει από τις περιγραφές αυτές στις περιπτώσεις που ορίζονται από το, κοινωτικό, από το εθνικό δίκαιο. Και βλέπουμε ότι στη νέα έκδοση του σχεδίου διαχείρισης το Μάρτιο του 2015, 2015 αφαιρέθηκε αυτή η προδιαγραφή και τέλος σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις ε, Σεπτεμβρίου του 1997 σε ό,τι αφορά Α, τα ζώα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Κεκτημένου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκ τούτου δεν είναι αρμόδια για την εφαρμογή τη Ευχαριστώ πολύ. Να ξαναξεκινήσω. Μιλήσατε με μεγάλη ταχύτητα καταρχήν. Υπάρχουν βουλευτές που θα ήθελαν το λόγο. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Γιάρ. Νομίζω ότι η δηλώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ε, επαρκής και ικανοποιητικές. Γι' αυτό θα πρότεινα να κλείσει αυτή η αναφορά. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω το εξή ότι έχουμε ένα, μια διαδικασία. Κλείνει η αναφορά και αν προκύψουν καινούργια τεκμήρια, ασφαλώ μπορεί να ξανανοίξει η αναφορά, αλλά προ το παρόν δεν επαρκεί η βάση των πληροφοριών, τα τεκμήρια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα για να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Προτείνω λοιπόν να κλείσει και να ενημερωθούμε στη συνέχεια. Σύμφωνα με τις ε, πληροφορίες θα κλείσουμε την αναφορά. Εάν ανακύψουν νέες πληροφορίες τότε θα το δούμε. Περνάμε στην επόμενη που είναι η 50 κάθετος 2015 ε, για την παράληψη εκπόνησης ε, στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης στην περιοχή Τόρε Γκράντε του Δήμου Οριστάνου. Έχει έρθει ο αναφέρον. Όχι, άρα δίνουμε το λόγο στη Μαγδαλένα Προύνα, στην Επιτροπή. Ναι, θα τα πω πιο αργά αυτή τη φορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη ρήπανση Οι διερμηνείς ζητούν να διαβάζετε αυτά που σας έχουν γράψει με όχι την ταχύτητα την προηγούμενη. Σε ό,τι αφορά τη ρήπανση λοιπόν του υπεδάφου, του πρώην βιομηχανικού εδάφου και από τι πληροφορίε που έχουμε λάβει από τον αναφέροντα, φαίνεται ότι οι δραστηριότητε εκαθάριση προβλέπονται όπω ε, βλέπει και η Ιταλική νομοθεσία, ή όπω συμπονήθηκα, σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη παραβίαση της οδηγίας, ε, της κοινωτικής οδηγίας, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι τα σχέδια για τη χρήση της γης που καθορίζουν τη χρήση τέτοιων μικρών εκτάσεων σε τοπικό επίπεδο και η ίσονο σημασία τροποποίησης ε, προϋποθέτουν και προαπαιτούν περιβαλλοντική μελέτη μόνο εφόσον υπάρχει ε, σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Αλλά μιας και η τροποποίηση της εγκατάστασης αφορά ένα έργο προς κατασκευή σε ε, οικιστική περιοχή, σε μια πρώην βιομηχανική περιοχή μόνο αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού. Δεν είναι σαφές από τις πληροφορίες που μας παρήχε ο αναφέρον. Με ποιο τρόπο λοιπόν αυτή η τροποποίηση ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και έτσι να προαπαιτεί τη διαδικασία SEA. Επιπλέον, από τις πληροφορίες που λάβαμε από τον αναφέροντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, βρήκε τεκμηρία για το ότι οι τοπικές αρχές ως τώρα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή της, του κανονισμού σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αυτή. Τέλος, ε, τα εθνικά διοικητικά όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που ήδη έχουν μεταφερθεί σε εθνική νομοθεσία είναι υπεύθυνα για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και έχουν τα παρετέντικα μέσα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αν όντω δικαιολογούνται οι ανησυχίες που εκφράζονται. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν παρεμβάσεις, παρακαλώ. Ο Πίτερ, έχετε το λόγο. Εγώ θεωρώ ότι η κατάσταση προσωμιάζει και αυτή που είχαμε και στην προηγούμενη φορά μικρές αλλαγές σε μια προστατευμόμενη περιοχή. Και οι τοπικές αρχές είναι αυτές που τελικά θα πρέπει να κρίνουν κατά πόσον υπάρχει πρόβλημα. Μετά από μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε τεκμήρια για παραβίαση της κοινωτικής νομοθεσίας. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ θα πρότεινα και αυτή να κλείσει η αναφορά, σε περίπτωση που προκύψουν εκ των υστέρων ε, άλλα στοιχεία και πληροφορίες οι οποίες ε, μας φέρουν σε κατάσταση αμφιβολίας, μπορούμε να ανοίξουμε την αναφορά. Αλλά στην παρούσα φάση θα έλεγα να την κλείσουμε την αναφορά. Ναι, πράγματι, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό αυτό. Κλείνει η αναφορά και αν ανακύψουν άλλες πληροφορίες, νέες πληροφορίες θα επανέλθουμε. Περνάμε στην αναφορά 1199-2011 που θα μας ε, παρουσιάσει ένας Ισπανός και άλλοι 16 αναφέρονται σε σχέση με την ε, παραβίαση ε, δικαιωμάτων ψήφου των απόδημων Ισπανών. Θα μας παρουσιάσει την αναφορά ο Γκαμπριέλ Τελακρούθ. Έχουμε δύο αναφέροντες που είναι ε, ε, παρόντες, ε, Μαρία Τελασνιέβες και Γκαμπριέλ Τελακρούθ. Μαρία Τελασνιέβες καταρχήν, έχετε το λόγο. Η αναφέρουσα έχει το λόγο. Ακούγεται. Εντάξει, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ που μας ε, καλέσατε όταν ε, συνέταξα αυτή την αναφορά δεν συμμετείχα σε τέτοιες δημοκρατικές διαδικασίες γιατί ε, μετέβη στη Φιλανδία 13 χρόνια πριν, εργάστηκα στο Πανεπιστήμιο το φιλανδικό κράτος ε, με πληρώνει, καταβάλει το μισθό μου και το 2010 άλλαξε ο νόμος με βάση ένα γραφειοκρατικό άχθος που υπάρχει και έτσι είναι δύσκολο να ασκήσω το, το δικαίωμα του εκλέγην. Όταν υπέβαλα αυτή την αναφορά, αυτό έγινε μετά τις ευρωεκλογές και με βάση αυτή τη μέθοδο θα πρέπει κανείς να ζητήσει να ασκήσει το δικαίωμά του. Ε, μετά θα πρέπει να περιμένει, να λάβει ένα δελτίο, να το ξανααποστείλει και να περιμένει το χρόνο των εκλογών και δυστυχώς ε, λαμβάνω πολύ αργά το ψηφοδέλτιό μου γιατί υπάρχουν διχογνωμίες ως προς τους υποψηφίους και περιμένω ε, δύο εβδομάδες μέχρι να λάβω τα ψηφοδέλτια. Στη δική μου περίπτωση από το 2010 δεν μπόρεσα να ασκήσω το δικαίωμα το εκλογικό δικαίωμα, γιατί αυτή η διαδικασία είναι πολύ σχηνοτενής. Στο Τολέδο, όταν κάλεσα τους αρμοδίους, μου είπαν ότι δεν έχει νόημα να κάνω καταγγελία εναντίον τους, αλλά θα πρέπει να κάνω καταγγελία στα ταχυδρομεία. Υπάρχουν δύο εκατομμύρια Ισπανοί που ζουν στο εξωτερικό και αυτή η διαδικασία ε, άσκησης του δικαιώματος ε, του εκλέγην έχει μία ανωδική πορεία και φτάνει από το 5% στο 32% και δεν φταίνε πάντα τα ταχυδρομεία. Καταρχήν αυτός ο νόμος ισχύει για να μην ε, γίνουν καταχρήσεις στην Νότια Αμερική. Υποτίθεται, εγώ ζω στην Ευρώπη και δεν θέλω να χάσω τα δικαιώματά μου ιδιαίτερα ως προς τη, συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Οι, οι εκλογές στην Ισπανία είναι πολύ σημαντικές για μένα, οι, μου ζουν στην Ισπανία. Εγώ θα ε, ξαναμετακομίσω στην Ισπανία, θα επιστρέψω στη χώρα μου μπορώ να ψηφίσω στις δημοτικές εκλογές στο Ελσίνκι, αλλά έχουν μεγάλη σημασία οι εθνικές εκλογές και οι ευρωεκλογές. Γιατί εντάξει, δεν πρέπει να γίνονται καταχρήσει στη Νότιο Αμερική, γιατί οι εκλογικοί κατάλογοι δεν ήταν σωστοί και δύο νεκροί υποτίθεται ότι άσκησαν το δικαίωμά τους, αλλά οι Ισπανικές αρχές δεν ε, έχουν τα κατάλληλα ε, μέσα να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα της απάτης στους εκλογικούς καταλόγους. Γι' αυτό οι, Ισπανοί, οι Ισπανικές αρχές πρέπει να λύσουν αυτό το θέμα σε επίπεδο εκλογικών ε, καταλόγων. Αυτό το σύστημα ε, χρησιμοποιήθηκε και πριν και το 2008 χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα για τοπικές εκλογές και τότε η ποσοστή αναλογία μειώθηκε, δηλαδή από 31,88% μειώθηκε το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματος γύρω στο 5%. Άρα δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα, αλλά μετά έγινε μία γραπτή σύσταση από την Εκλογική Επιτροπή που ακριβώς αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν μπορούν οι πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Αυτό το σύστημα εισήχθη επίσημα το 2010 και μειώθηκε η συμμετοχή στις εκλογές από 32% σε 5%. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει αυτό το θέμα. Εγώ, εγώ είμαι ε, Ισπανός πολίτης, ζω στη Φιλανδία και πιστεύω ότι επειδή ασκώ το επάγγελμά μου στη Φιλανδία, στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχω τη δυνατότητα να ασκώ το δικαίωμα του εκλέγην. Είμαστε δύο εκατομμύρια που ζούμε στο εξωτερικό. Μιλώ για Ισπανούς. Δεν ξέρω πόσοι ζουν στην Ευρώπη, αλλά οι περισσότεροι ζούμε στην Ευρώπη και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση κάπως. Γιατί οι Ισπανικές αρχές ε, δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα, το αγνοούν. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορούσα να σας μιλήσω για πολιτικές ευθύνες, Και αν σκεφτούμε τι επέλυσε αυτός ο νόμος, τι πέτυχε, το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο. Το 2008 η εκλογική επιτροπή μίλησε για 0,44% επιστροφών των ψηφοδελτίων. Γιατί αυτοί που θα ασκούσαν το δικαίωμά τους θα στην ουσία είχαν αποβιώσει. Γι' αυτό θα πρέπει να επιληθεί το θέμα των εκλογικών καταλόγων. Το θέμα δεν είναι μόνο τοπικό. Δηλαδή να αφορά τους κατοίκους εξωτερικού αλλά και εσωτερικού. Σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, δεν μπορούσα να ελέγξω το χρόνο μου. Η Μόνικα θα ήθελε να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα μόνο να πω ότι από τότε που άρχισε να ισχύει αυτός ο νόμος Θεωρώ ότι έχει υπάρξει καταστρατήγηση της αρχής ισότητας των πολιτών, η οποία όμως κατοχυρώνεται από το Ισπανικό Σύνταγμα, διότι έχει δυσχερανθεί η θέση των Ισπανών που ζουν στο εξωτερικό και έχουν δυσκολευτεί στην προσπάθειά τους να ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά αν το Ισπανικό κράτος δεν προσπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών του, των υπηκόων του, εμείς είμαστε Ισπανοί πολίτες παρόλο που ζούμε στο εξωτερικό, ε, τότε προσφεύγουμε σε ανώτερα θεσμικά όργανα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρέμβει σε ένα θέμα εργατικού δικαίου στην Ισπανία και τελικά αυτό επηρέασε το ψήφισμα που υπήρξε για τον έλεγχο της προσωρινής εργασίας και των προσωρινών συμβάσεων. Αφού το έκανε σε αυτό το τομέα θεωρώ ότι θα μπορούσε να παρέμβει και στο δικό μας ε, θέμα και ότι έχει αρμοδιότητα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ να δώσουμε το λόγο στη Μόνικα, μέλος της ε, Επιτροπής της Σχετικής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καταρχάς, Η Επιτροπή θεωρεί ότι όντω είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί κανείς να συμμετάσχει στις εκλογές, ότι έχει το δικαίωμα ο πολίτης να ψηφίσει και να ασκήσει το δημοκρατικό του δικαίωμα συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία παρόλο, παρόλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα ε, αρμοδιοτήτων και κατανομής αρμοδιοτήτων. Ε, δυσκολευόμαστε να παρέμβουμε σε θέματα εκλογών. Έχουμε εξουσία και αρμοδιότητα να παρέμβουμε για τη διοργάνωση των ευρωεκλογών και των τοπικών εκλογών, τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά όχι σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Από τη στιγμή που το κράτος το εκάστοτο εγγυάται τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές, έχουμε το νόμο 76, τότε έχει την αρμοδιότητα το κράτος μέλος να διοργανώσει τις εθνικές εκλογές με τον τρόπο που επιθυμεί. Επομένως δυσκολευόμαστε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει καταστρατήγηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω την προσοχή στο νέο νομοσχέδιο για κοινοβουλευτικές εκλογές, στο νέο κανονισμό, το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και με την υιοθέτηση ε, αυτού του κειμένου ελπίζουμε ότι θα μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τη δημοκρατική διαδικασία του εκλέγην στις ευρωπαϊκές εκλογές, στις ευρωεκλογές, να διευκολυνθεί αυτό και έτσι να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που έχουν συναντήσει οι πολίτες και να μπορέσουν να συμμετάσχουν πιο απρόσκοπτα στις ε, εκλογές του 2019. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ σειρά των βουλευτών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους αναφέροντες, όχι μόνο για την παρουσία τους, αλλά διότι μας εξήγησαν με πολύ συνοπτικό και συγκεκριμένο τρόπο ε, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βιώνουν. Και θα ήθελα καταρχάς να σας ε, επισημάνω, παρακαλώ ησυχία, θα ήθελα να σας ε, επισημάνω πόσο ονομάζεται αυτή η ψηφοφορία στην Ισπανία. Είναι παρακλητή ψήφος, θα πρέπει κανείς να παρακαλέσει γι' αυτό. Είναι ένα δικαίωμα του πολίτη, όμως συγκεκριμένοι πολίτες που ζουν εκτός της χώρας, αλλά είναι Ευρωπαίοι πολίτες και ζουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, είναι ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να παρακαλέσουν, να ζητήσουν για να το έχουν και θα πρέπει αυτοί να ασχοληθούν για να το διαχειριστούν και να μπορούν να το ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Και αυτό υπάρχει στην Ισπανία από το 2010 ε, δικαίωμα να εκλέγουν είναι ε, οι Ισπανοί που μένουν στην Ισπανία και όσοι Ισπανοί μένουν εκτός Ισπανίας πρέπει να το ζητήσουν αυτό το δικαίωμα, γι' αυτό και το ονομάζουμε παρακλήτο δεν έχουν ε, διορθωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι και γι' αυτό έχουν υπάρξει διάφορα προβλήματα και γι' αυτό έχει γίνει πιο δυσχερής η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των Ισπανών που ζουν στο εξωτερικό, εκτός Ισπανίας. Το ξέραμε αυτό. Δεν είναι θετική έκβαση λοιπόν. Θα ήθελα όμως να τονίσω και να υπογραμμίσω το ότι το εξής. Η Επιτροπή προφανώς αναγνωρίζει ότι η αρμοδιότητα για την εκλογική νομοθεσία στις εθνικές εκλογές έχουν αποκλειστικά και μόνο τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι σαφές. Όμως κάτι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τις Ισπανικές Αρχές. Σίγουρα με τη νέα νομοθεσία που ε, και τον νέο κανονισμό που εξετάζεται στην Ευρώπη για τη ρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας έχετε έρθει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς στα κράτη-μέλη και άρα με τους Ισπανικούς αρμόδιους φορείς. Επομένως, Ξέρετε ότι η Ισπανία θα ήθελε η Ισπανία εκτός της χώρας να ψηφίζουν απρόσκοπτα, αλλά δεν έχει τη τεχνογνωσία για να τους διευκολύνει απολύτως 100% σε αυτό το εγχείρημα. Και μπορείτε να τους βοηθήσετε η γραφειοκρατική διαδικασία, τα έξοδα, ο χρόνος και το αίσθημα της ματέωσης που βιώνει ο Ισπανός πολίτης που ζει στο εξωτερικό είναι οι αιτίες για τις οποίες τελικά καταμετρώνται πολύ λίγες ψήφοι Ισπανών του εξωτερικού. Στη, σήμερα, στην εποχή που ζούμε, με την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας, με το ότι είναι τόσο ε, εύκολο να περάσουμε τα σύνορα, γιατί δεν έχουμε σύνορα ούτε ε, απτά, ούτε οικονομικά, ούτε καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρίμα να πρέπει να χρησιμοποιούμε αναλογικά μέσα για κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνεται απρόσκοπτα και εύκολα με τις εφαρμογές της τηλεματικής. Και για να κλείσω, για να δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους συναδέλφους, να πω ότι στις εκλογές του 2008 και τις τελευταίες ε, ε, εκλογές του Δεκεμβρίου 2015 μειώθηκε τέσσερις φορές, υποτετραπλασιάστηκε η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των Ισπανών του εξωτερικού. Ε, περίπου 7% μόνο από αυτούς που το ζήτησαν μπόρεσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενώ ο ισπανικός πληθυσμός που έχει μετικήσει και έχει φύγει εκτός των ισπανικών συνόρων έχει αυξηθεί δραματικά πάνω από 2 εκατομμύρια και φέτος μόνο 60.000 άνθρωποι. Είναι προβλήματα που δεν επηρεάζουν μόνο το Ισπανικό κράτος. Η έλλειψη ομοιομορφίας στις απαιτήσει και ε, σε αυτά που πρέπει να εκπληρώσουν ως διαδικαστικά ε, προαπαιτούμενα οι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό προκειμένου να ψηφίσουν υπάρχουν παντού. Κάποιοι Ευρωπαίοι πολίτες το βρίσκουν πιο εύκολο να ψηφίσουν σε διάφορες διαδικασίες και κάποιοι λιγότερο στις ίδιες εκλογικές διαδικασίες. Επομένως, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το περσινό προτείνει να έχουμε την επιστολική ψήφο, να έχουμε την ψήφο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω διαφόρων ψηφιακών μέσων, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο πολίτης και τουλάχιστον στις ευρωεκλογές να μπορέσουμε να ε, κάνουμε απολύτως ομοιόμορφο τον τρόπο εκλογικής διαδικασίας. Από τη στιγμή που υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία, θεωρούμε ότι υπάρχει καταστρατήγηση του δικαιώματος αυτού για τους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Το να μπορέσει κανείς να ψηφίσει από το εξωτερικό ουσιαστικά είναι ένας δρόμος μετεμποδίων και πρέπει να είμαστε ικανοί να βελτιώσουμε τους τρόπους με τον οποίο ασκεί κανείς το εκλογικό του δικαίωμα. Και προτείνω τα εξή. Από την Επιτροπή των Αναφορών, εμείς να στείλουμε επιστολή στις Ισπανικές Αρχές, να εκφράζουμε την ανησυχία που έχουμε για αυτό το θέμα και να ζητούμε την υιοθέτηση των απαραίτητων μέτρων για να εγγυηθεί το Ισπανικό κράτο, στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στους Ισπανούς πολίτες που ζουν στο εξωτερικό με βάση την Ισπανική νομοθεσία του 2010 έτσι όπως έχει ψηφιστεί και εγκριθεί. Νομίζω ότι είναι κάτι το απλό, το συνοπτικό, το συγκεκριμένο και το περιεκτικό και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε επαφή με τα κράτη-μέλη και άρα και με την Ισπανία και να επαληθεύσει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα από την τελευταία φορά που ήρθαν σε επαφή κυρίως ό,τι αφορά την εφαρμογή του ψηφίσματος για την ε, εκλογική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος, επόμενη ομιλήτρια έχει το λόγο. Καλημέρα σας και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για την παρουσίαση ε, των αναφορών τους, για όλη αυτή τη δουλειά, για όλο αυτό το έργο κινητοποίησης το οποίο έχουν ε, επιτελέσει. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα παράπονα που έχει λάβει η Επιτροπή μας είναι πολύ άριθμα σε ό,τι αφορά την καταστρατήγηση του δικαιώματος ε, συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλές από αυτές τις αναφορές αφορούν τη δική μας χώρα, την Ισπανία, πόσο μάλλον μετά τη μεταρρύθμιση του ε, εκλογικού νόμου του 2010, εκλογικός νόμος ο οποίος ε, επιβάλλει τον, την παρακλητή ψήφο την οποία εμείς ε, λόγω συνήχησης και παρήχησης ονομάζουμε συχνά κλεμμένη ψήφο γιατί τελικά στερεί από το δικαίωμα να ψηφίσουν πάνω από, στερεί πάνω από το 70% των Ισπανών που ζουν στο εξωτερικό από το δικαίωμά τους τελικά να ψηφίσουν γιατί υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια και ο Υπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος Φερνάντο Δία είχε αναγνωρίσει ότι πρέπει να το κοιτάξει το θέμα γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να ψηφίσει κανείς από το εξωτερικό. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται για στέρηση βασικού ε, δικαιώματος και για χειραγώγηση του εκλογικού αποτελέσματος. Μιλούμε για 2 εκατομμύρια Ισπανούς που ζουν εκτός της επικράτειας και 2 εκατομμύρια ψήφοι οι οποίες χάνονται. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο Κατανοούμε όλοι ορισμένες κυβερνήσεις λόγω κρίσης, επειδή οι άνθρωποι πρέπει να μετικήσουν, ε, καταλαβαίνουν ορισμένες κυβερνήσεις ενδεχομένω να, να μην θέλουν τόσο εύκολα να μπορούν να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε ένα νομοσχέδιο με μια νομοθεσία που να εγγυάται το δικαίωμα ψήφου στους Ισπανούς του εξωτερικού με ισότιμο τρόπο σε σχέση με τους κατοίκους εντός της χώρας. Βεβαίως, επανειλημμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αυτή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και το δέχομαι. Ωστόσο, το άρθρο 10, δάφιο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με το πιο ανοιχτό δυνατό τρόπο και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη σε ό,τι αφορά το επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται. Με βάση αυτό, με βάση αυτό το εδάφιο, ε, το περιεχόμενο του εδαφίου δεν γίνεται σεβαστό στην Ισπανία γιατί έχουμε καταστρατηγήσει παραβίαση αυτού του δικαιώματο για εκατοντάδε. χιλιάδες, δύο εκατομμύρια σα λέω, Ισπανούς πολίτες που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και που ζουν στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι είναι ξεκατάφορη η καταστρατήγηση του δικαιώματος ε, για την ελεύθερη κυκλοφορία και κατοικία παραμονή ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό επίσης κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 45 της Ευρωπαϊκής Χάρτας ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επιθυμούμε να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά. Συμφωνούμε απολύτως με την σύνταξη επιστολής στις Ισπανικές Αρχές που θα εκφράσει την ανησυχία της Επιτροπής Αναφορών σε σχέση με αυτό το ζήτημα και προτείνουμε ε, μια πρωτοβουλία παρακολούθησης της υπόθεσης και συνεδρίαση με συμμετοχή μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων έτσι ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για το τι γίνεται στην πράξη ε, στα διάφορα κράτη-μέλη για την ε, ψήφο ε, από το εξωτερικό και θέλουμε και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΑΦΚΟ να επιληφθεί του θέματος και να συνεργαστεί με την Επιτροπή Αναφορών και να ασχοληθεί όχι μόνο με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τη συνταγματική σκοπιά, αλλά και με την ύπαρξη διακρίσεων ε, των μεν και των δε, ε, κάτι το οποίο αναφέρεται σε όλες αυτές τις αναφορές που μας έχουν υποβληθεί. Σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στους αναφέροντες, ελπίζουμε να διατηρηθούν ανοιχτέ αυτές οι αναφορές και να υπάρξει μια πιο συγκεκριμένη έκβαση ε, της συνέχειας που θα δοθεί σε αυτές τις αναφορές στις επόμενες συνεδριάσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα όσα προελέχθησαν γιατί στην η οικογένειά μου είναι, είμαι η μόνη που δεν έχω ισπανική ηθαγένεια. Τα παιδιά μου μπορούν να ψηφίσουν στην Ισπανία, αλλά δεν άσκησαν αυτό το δικαίωμα ποτέ. Άρα μιλάμε για την αναθεώρηση του νόμου, γιατί δυστυχώς τα ψηφοδέλτια δεν έφταναν στο χρόνο που έπρεπε και δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν τώρα με τη νέα νομοθεσία φτάνουν τα έγγραφα αλλά στο ίσα ίσα για να μπορέσουν να μπουν στο διαδίκτυο, να εγγραφούν και ούτω καθεξής. Τις τελευταίες ε, μέρες όμως καταλαβαίνετε υπάρχει κορεσμός ε, του διαδικτύου και δεν μπορούν να εγγραφούν εγκαίρους. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί συνέχεια όπως πρότειναν πολύ. Κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν μπορεί τόσοι άνθρωποι στο εξωτερικό να μην μπορούν να ψηφίσουν. Το θυμάμαι γενικότερα και ο πατέρας τους πολλές φορές ήθελε να ψηφίσει αλλά τα ψηφοδέλτια έφταναν μία εβδομάδα μετά τις εκλογές. Δηλαδή θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, να βρεθεί μία λύση. Η Σολεντάτ Καμπεθόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η μεταρρύθμιση της παρακλητικής άσκησης του δικαιώματος του εκλέγην δεν λειτουργήσε σωστά αυτό. Το αναγνώρισαν και οι σοσιαλιστές και στην ε, προεκλογική τους εκστρατεία τόνισαν ότι θα επιλύσουν αυτό το θέμα της ε, παρακλητικής άσκησης του δικαιώματος και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσει για να μπορέσουν οι Ισπανοί οι να μπορέσουν να ψηφίσουν και στο εξωτερικό και είχαμε μιλήσει για παρεκκλήσεις στο αρχικό μας πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εγγύηση άσκησης αυτού του δικαιώματος του εκλέγην από εκείνους που έχουν το δικαίωμα άσκησής τους. Φυσικά δεν θέλουμε να υπάρξει ε, αποφυγή ασκήσεως ή παρακόλληση ασκήσεως αυτού του δικαιώματος. Όμως επειδή υπάρχουν δυσκολίες είναι δύσκολο να επικαιροποιηθεί ο εκλογικός κατάλογος των ε, πολιτών που ζουν στο εξωτερικό. Και Γι' αυτό ακριβώς είναι δύσκολο να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα του εκλέγην. Γι' αυτό προβάλλουμε αυτή τη μεταρρύθμιση έτσι ώστε να ασκηθεί πλήρως το δικαίωμα του εκλέγην από τους Ισπανούς υπηκόους που διαβιούν στο εξωτερικό και να υπάρχει πλήρης αντιστήχηση του εκλογικού σώματος και των εκλογικών ε, καταλόγων. Βεβαίως, η κάτοικοι είναι πάρα πολύ και μιλάμε για μείωση της άσκησης του δικαιώματος από το 32% στο 5%. Δηλαδή μιλάμε για μία μείωση της άσκησης του δικαιώματος της τάξης περίπου του 25-26%. Πρόκειται λοιπόν για ένα γραφειοκρατικό πρόσκομα που είναι ύψη της σημασίας. Με αυτή τη νέα μεταρρύθμιση πιστεύουμε ότι θα λυθεί εν μέρη το ζήτημα. Το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματος του εκλέγην είναι ύψης της σημασίας και πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση δεν ήταν η βέλτιστη δυνατή, αλλά υπάρχει η εγγύηση του δικαιώματος, της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγην και στο εξωτερικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως θα πρέπει να βελτιώσουμε το πλαίσιο για τους ε, κατοίκους σε άλλες χώρες, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, Σολεδάδ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο θεωρούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει λίγο να τα βάλουμε σε μια σωστή νομική βάση. Υπάρχει το άρθρο 223 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει σχέδιο για τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων με στόχο την εκλογή των μελών του κατά ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη-μέλη ή σύμφωνα με κοινέ αρχές όλων των κρατών μελών. Εδώ είναι η βάση. Δηλαδή, και αυτό εν συνεχεία αποφασίζεται από το Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί ε, με μια συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία και από το Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια απόφαση από τη συνθήκη ότι η εκλογή θα γίνεται με ενιαία διαδικασία και με κοινέ αρχές. Επομένως, καταρχάς η αρμοδιότητα είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άσχετα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καταλήξει σε μια ενιαία εκλογική νομοθεσία διότι δεν τα βρίσκει το Συμβούλιο και δεν τα βρίσκουν τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η βάση. Και ακριβώς επειδή δεν μπορούν να τα βρουν, φτιάχνουν μερικές γενικές αρχές και τα υπόλοιπα τα αφήνουν να τα ρυθμίσει η Εθνική Εκλογική Νομοθεσία. Θα σας πω λοιπόν αυτό το θέμα το οποίο το έχω θέσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πριν εκλεγώ ως Ευρωβουλευτής, γιατί ακούστε τι πρόβλημα υπάρχει με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Σε όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από τη Λετωνία και την Ελλάδα, προκειμένου ένας βουλευτής Εθνικού Κοινοβουλίου να είναι υποψήφιος για Ευρωβουλευτής, μόνο στην Ελλάδα και στη Λετωνία πρέπει πρώτα να παρετηθεί από βουλευτής για να έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής. Ενώ σε όλα τα κράτη-μέλη τα υπόλοιπα μπορείς να είσαι βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου, να κατέβεις στις ευρωεκλογέ και αν εκλεγείς στο Ευρωκοινοβούλιο διαλέγεις ανάμεσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο στην Ελλάδα επιβάλλεται αυτή η ρύθμιση και στη Λετωνία. Και εγώ προσωπικά και άλλοι πέντε συνάδελφοι παρετηθήκαμε από βουλευτές προκειμένου να έχουμε το δικαίωμα να είμαστε υποψήφοι αυτό είχα εξηγήσει ότι είναι αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διότι δημιουργεί διακρίσει σε σχέση με το πώ εκλέγεστε εσεί οι υπόλοιποι. Αν κάποιο από εσά ήταν μέλο Εθνικού Κοινοβουλίου, είχε δικαίωμα να είναι υποψήφιο και αν εκλεγόταν θα διάλεγε ανάμεσα στα δύο κοινοβούλια. Εγώ και άλλοι πέντε συνάδελφοι που έχουμε έρθει από την Ελλάδα παρετηθήκαμε και δεν γνωρίζαμε αν θα εκλεγούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είχα πει τότε ότι αυτό είναι παράνομο. Άρα λοιπόν υπάρχουν κατά την άποψή μου μερικές γενικές αρχές οι οποίες πρέπει να τηρούνται παντού. Και μία από τις γενικές αρχές φυσικά έχει σχέση και με τον τρόπο συμμετοχής, δηλαδή με το εκλέγην των πολιτών οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την αίτηση των Ισπανών. Διότι πρέπει να είναι έτσι η ρύθμιση της εθνικής νομοθεσίας που να μην δημιουργεί διακρίσεις, να μην παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο και είναι παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν σε διευκολύνει να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα διότι βρίσκεσαι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας ασκήσει δικαίωμα ευρωπαϊκό, δηλαδή το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης. Επομένως, αν αποδειχθεί ότι καταστρατηγείται αυτό από κάποιο κράτος μέλος και εν προκειμένου από την Ισπανία σημαίνει ότι παραβιάζεται εν προκειμένου το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαίνει ότι η Κομισιόν πρέπει να πάρει μέτρα ούτως ώστε να συμμορφωθεί η Ισπανία με τη ρύθμιση αυτή. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες να δούμε για ποιο λόγο στην Ισπανία γίνεται αυτή η κατάσταση. Θα σας πω τι γίνεται με την Ελλάδα, γιατί έχουμε και εμείς πολλού Έλληνες. Υπάρχει δυνατότητα Έλληνες που κατοικούν στο Βέλγιο αυτοί είτε μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους του Βελγίου και να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ, αλλά ψηφοδέλτια βέλγικα, είτε να εγγραφούν έγκαιρα στους εκλογικούς καταλόγους στην Ελλάδα, όσοι επιθυμούν, και να ψηφίσουν στην, στο Βέλγιο ψηφοδέλτια ελληνικά και πηγαίνουν και ψηφίζουν στην πρεσβεία που υπάρχει εδώ στο Βέλγιο, στην ελληνική πρεσβεία. Αυτό γίνεται σε όλα τα μέρη Τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του Έλληνε πολίτε. Και μέχρι στιγμή, τουλάχιστον εμεί στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα παραδόξω δεν έχουμε πρόβλημα. Και υπάρχει ομαλή διαδικασία. Άρα θεωρώ ότι εφόσον αυτό μπορεί και το κάνει η Ελλάδα, προφανώ θα μπορούσε να το κάνει και η Ισπανία. Είναι θέμα λοιπόν διοικητική ρύθμιση και πολιτική απόφαση. Αν λοιπόν στι τεχνικέ λεπτομέρειε αποδεικνύεται ότι το Ισπανικό κράτο για κάποιου ειδικού λόγου κολλησιεργεί δεν φτιάχνει τους εκλογικούς καταλόγους και στο τέλος δημιουργεί πρόβλημα και οδηγεί σε αυτή την παρακλητική ψήφο όπως την είπατε, τότε υπάρχει αρμοδιότητα της Επιτροπής, υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά η Κομισιόν για ενδεχόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών στην Ισπανία. Θα το δούει όμως αυτό η Κομισιόν με βάση τις λεπτομέρειες. Για ποιο λόγο στην Ισπανία δεν μπορεί να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των εκλογικών καταλόγων, εφόσον ξέρουμε πότε θα γίνουν ευρωεκλογέ, θα γίνουν το 2019 το Μάιο. Προφανώς θα μπορούσαν οι εκλογικοί κατάλογοι να κλείσουν το Φεβρουάριο του 2019. Μέχρι τότε όσοι είναι μέχρι το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο του 19 που ζουν σε άλλες χώρες να εγγραφούν στους καταλόγους και βεβαίω σε συγκεκριμένους χώρους ή στην πρεσβεία της Ισπανίας λέμε στο Βέλγιο ή σε άλλους χώρους να γίνουν οι εκλογές. Άρα κάτι άλλο υπάρχει. Και αυτό το άλλο ενδεχόμενα μπορεί να είναι μια πολιτική απόφαση του Ισπανικού κράτους να αποκλείσει όσους έχουν πάει στο εξωτερικό γιατί προφανώς θα ψηφίσουν με ένα διαφορετικό κριτήριο. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή η υπόθεση αυτή, να μας απασχολήσει σοβαρά, διότι δεν αφορά μόνο την Ισπανία, αφορά το δικαίωμα εκλέγεστε και εκλέγειν. Ένα, το παράδειγμα που σας έφερα από την Ελλάδα δείχνει ότι έχουμε πολλές πλευρές να εξετάσουμε, άρα να συγχαρώ τους συναδέλφους που έθεσαν το θέμα τους petitioners και να αφήσουμε ανοιχτή την υπόθεση, να δούμε πώς θα πάμε παραπέρα και συμφωνώ με τις εισηγήσεις των συναδέλφων από την Ισπανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής. Sí, gracias. Bueno, a ver si... Ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση. Δεν μιλάμε μόνο για τις ευρωεκλογέ. έτσι δεν είναι. Ωραία, για να είμαι σίγουρος για τι πράγμα μιλάμε. Χαίρομαι για την παρέμβαση ε, του κυρίου Μαριά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του ζητήματος. Εάν ένα τόσο θεμελιώδης ε, δικαίωμα παραβιάζεται, όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων, από τις ε, εθνικές ε, νομοθεσίες. Αυτό θα πρέπει να αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων και ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το διευθετήσει η ΠΕΤΗ το ζήτημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες πραγματικά με συγκινούν γιατί ενδιαφέρονται στην τήρηση των δικαιωμάτων τους, το σεβασμό των δικαιωμάτων και μιλούν για μία ευνομούμενη κοινωνία την οποία προωθούν με αυτό το μέσον. Δηλαδή χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους έτσι ώστε να εκθέσουν μία κατάσταση που αφορά θεμελιώδη παραβίαση άσκησης ενός δικαιώματος μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής μας ε, κοινωνίας. Πέρα λοιπόν από το θαυμασμό μου θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα ζωτικής σημασίας. Μιλάμε για δύο πτυχές όμως παράλληλα που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά αφορούν διαφορετικές καταστάσεις. Μιλάμε για ένα καυκικό σενάριο καταρχήν, όπου η θέση σε εφαρμογή του νόμου από τις δημόσιες αρχές έχει καταστροφικό αποτέλεσμα, δηλαδή υπάρχει κόλληση μια σχηνοτενής διαδικασία και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα, αλλά ε, μόνο αν υπάρχει δόλος πραγματικός που δεν συμφωνώ ε, με το συνάδελφο Καμπεθόν, δεν νομίζω ότι υπήρχε δόλος για την τακτική αυτή. Απλώς έχουμε να κάνουμε με ένα καυκικό σενάριο, δηλαδή ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής ή ο συνήγορος του πολίτη θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, δηλαδή όταν πλήττονται αυτά τα δικαιώματα. Τώρα, το δεύτερο θέμα που είναι η ο συνηγορος του πολιτη θα επρεπε να ασχοληθει με αυτο το θεμα δηλαδη οταν πληττονται αυτα τα δικαιωματα τωρα το δευτερο θεμα που ειναι η της σημασίας αφορά την παρακλητική ψήφο, που στο παρελθόν δεν υπήρχε στην Ισπανία. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, δεν μπαίνω σε μικροαψιμαχίες, δεν ανήκω πουθενά, είμαι ανεξάρτητος και δεν υπερασπίζομαι κανέναν, διότι την τελευταία 20 ετία οι κυβερνήσεις μας έφεραν καταστροφικά αποτελέσματα. Όμως η παρακλητική ψήφος στην περίπτωση της ε, Ισπανίας κάνει μία διάκριση μεταξύ πολιτών. Δηλαδή για τους μεν θα πρέπει να υπάρχει παράκληση, δηλαδή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να εκφράσουν καταρχήν το ενδιαφέρον συμμετοχής. Αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί γιατί και η ίδια η έννοια, η ενιολογική βάση αποτελεί πρόσκομα το οποίο δεν προϋπήρχε. Η μητέρα μου είναι Γαλλίδα και την καλούν από το προξενείο για να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει στον εκλογικό κατάλογο και στη συνέχεια ασκεί το δικαιωμά Δεν πρέπει να ζητήσει τίποτα ως γαλίδα υπήκος μπορεί να ψηφίσει. Δεν τη ζητείτε τίποτα. Αυτό το πρόσκομα λοιπόν, το επιπρόσθετο πρόσκομα είναι πολύ σοβαρό. Θεωρώ ότι η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Η Πέτη θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια μέσω εμπειρογνωμόνων να λήξει αυτή η πρακτική σε ολόκληρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για κατό, για κακό σημάδι όταν κάποιος πρέπει να εκδηλώσει εκ των προτέρων το ενδιαφέρον του, ότι πρέπει και ότι θέλει να ασκήσει ένα δικαίωμα. Το είπαν και πολλοί ε, προλαλήσαντες. Είναι δηλαδή μια επιπρόσθετη παράτυπη διαδικασία. Ελέγχ ότι η νέα κυβέρνηση θα αλλάξει τα πράγματα. Αλλά η Πέτη γιατί δεν αποστέλει μία επιστολή στο Ισπανικό Κοινοβούλιο προτρέποντας αυτή τη μεταρρύθμιση και αυτό να γίνει εξ ονόματος της Πέτη, όχι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει αν είναι δύο εκατομμύρια και ένας να ήταν, και ένας να ήταν, το δικαίωμα αυτό υπάρχει. Και είναι ιερό αυτό το δικαίωμα, να ασκήσει ο κάθε πολίτης αυτό το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Γιατί ε, δεν ξέρουμε πόσοι θα ψηφίσουν, ξέρουμε όμως ότι παρακολύονται από την ε, άσκηση αυτού του δικαιώματος. Ευχαριστούμε Ρίκε, ο Πίτερ Γιάρ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να δώσω λίγη κάπως αισιοδοξία προς το αναφέροντα. Χαιρόμαστε που κατέθεσε την αναφορά αυτή και πρόκειται πραγματικά για μια α, ιστορία επιτυχίας, ένα επίτευγμα της ενιαίας αγοράς Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ένα Ισπανό εργάζεται στην Γερμανία και το αντίστροφο είναι το κανονικό, αυτό που πρέπει να γίνεται, αυτό που επιθυμούμε, το ευκταίο. Και επίσης να πω ότι δεν είσαστε και οι μόνοι. Έχουμε και άλλα κράτη και άλλα κράτη και άλλες χώρες ε, που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και η Μεγάλη Βρετανία κατέθεσε μια σχετική αναφορά και αυτό έτσι να σα δώσει θάρρος φυσικά αποτελεί πρόβλημα. Γιατί το εκλογικό δικαίωμα είναι ένα βασικό θεμελιώδης δικαίωμα δημοκρατικό και δικαίωμα. Είχαμε και το σκάνδαλο που ψηφίζουν σε διάφορες περιπτώσεις πιο λίγοι πολίτες από ό,τι θα έπρεπε και αυτό δεν επιτρέπεται. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια γραφειοκρατία, αλλά δεν είναι δυνατόν η γραφειοκρατία να παρεμποδίζει το δικαίωμα από την ψήφο. Το τρίτο στοιχείο. Θεωρώ ε, ότι θα πρέπει να δώσουμε και μια αισιόδοξη νότα, κατεφετικό, από το τι ζητάμε. Αναφέρθηκε ότι το Κοινοβούλιο αναθεωρεί το εκλογικό δίκαιο και η Ισπανική κυβέρνηση διαπίστωσε το πρόβλημα και το αναγνώρισε. Είναι καλό αυτό. Είναι φετική είδηση. Δεν είναι σαν να αγνοούμε όλοι τον αναφέροντα. Όχι, ο αναφέρον αναγνωρίζεται από πολιτικής άποψης και νομοθετικός πώς έχουν κινητοποιηθεί τα πράγματα. Αυτό είναι καλό. Τώρα, ως Επιτροπή Αναφορών, τι πρέπει να κάνουμε. Είναι αδιαμφισβητητό ότι το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό με τις άλλες αναφορές για το εκλογικό δίκαιο, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η Ισπανία θα πρέπει και η Επιτροπή Νομοτικών Υποθέσεων να κοιτάξει τα θέματα αναθεώρηση του εκλογικού δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να υπάρχουν και κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για το, εκλογικό, το ευρωπαϊκό εκλογικό δίκαιο και το εθνικό εκλογικό δίκαιο. Αλλά υπάρχουν λοιπόν οι αρμόδιες επιτροπές και οι εμπειρογνώμονες και θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για αλλαγή. Αυτό που είναι επίσης αντιαμφισβήτητο είναι το ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε την ε, Ισπανική κυβέρνηση για την αναφορά με τη θετική έννοια. Ότι κοιτάξτε, ακούσαμε ότι θέλετε να αλλάξετε το εκλογικό δίκαιο. Σα παρακαλώ, λάβετε υπόψη και αυτό το πρόβλημα το υπάρχει και βρείτε μία λύση για του Ευρωπαίου πολίτε για να μπορούν να ασκούν το δικαίωμά του. Εκεί που αμφιβάλλω είναι στο τρίτο συμπέρασμα. Μπορεί να κλείσουμε την ε, αναφορά εφόσον αποστείλουμε την επιστολή προς την Ισπανική κυβέρνηση και παραπέμψουμε το θέμα στην αρμόδια επιτροπή. Μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση ή μπορούμε να την αφήσουμε ακόμα ανοιχτή την αναφορά. Εγώ θα ήμουν υπέρ του να την κλείσουμε την ε, αναφορά. Αλλά φυσικά μπορούμε να το συζητήσουμε και στην Επιτροπή. Ευχαριστούμε εκ νέου και τον ε, αναφέροντα. Και παρακαλώ όταν θα γυρίσετε στην πατρίδα σας να έχετε υπόψη και να το μεταβιβάσετε αυτό ότι το συνειδητοποιούμε ως βουλευτές το πρόβλημα της Επιτροπής Αναφορών ε, και ότι αυτό που αναφορά μόνο την Ισπανία αποτελεί ένα γενικότερο πρόβλημα και ίσως να αποτελεί αυτό ένα μικρό αν θέλετε ε, πρόβλημα της ενιαίας αγοράς και ως Ευρωκοινοβουλίο έχουμε την, ε, το καθήκον να το ρυθμίσουμε για να είναι αρμονικά τα πράγματα για τους πολίτες ήθελα να κάνω μία μικρή παρέμβαση όχι ως πρόεδρος αλλά ως Ισπανίδα Ευρωβουλευτής. Δέχομαι αυτά που είπε και η Σολεδά και ξέρουμε ότι ανέκυψαν, έγιναν και απάτες στις Βαλεαρίδες και γι' αυτό ακριβώς ελέγχθη ότι η έλεγχη δεν ήταν ε, επαρκείς γι' αυτό. Η Ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους, όμως η διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί και όταν ε, τέθη σε εφαρμογή αν και το κατά 75% είναι μία δωρεάν διαδικασία σε 17 χώρες, σε άλλες χώρες όχι, Υπάρχει και ένα θέμα με τις προθεσμίες, αλλά καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εγγύηση της άσκησης του δικαιώματος και μπορεί να βελτιωθεί φυσικά η διαδικασία. Ευπρόσδεκτη λοιπόν η αναφορά γιατί ό,τι μπορεί να βελτιωθεί ως προς τις προθεσμίες, την ευελιξία της διαδικασίας, Όλα αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Είναι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν. Ε, όταν άλλοι πολίτες μεταβαίνουν σε άλλη χώρα δεν μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, ενώ στην Ισπανία γίνεται κάτι τέτοιο. Επανέρχομαι ως πρόεδρος τώρα. Ναι, ναι, ναι, οι αναφέροντες μπορούν να λάβουν το λόγο πριν υποβάλω την ε, τελική μου πρόταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν έχω και τίποτα ιδιαίτερο να προσθέσω στην παρούσα φάση. Θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω την τοποθέτησή μου. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι τόσο διοικητική φύσεως. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, θεωρώ. Θεωρώ ότι είμαστε πλέον αρκετά εμπειροί για να κατανοούμε ότι η μέθοδος δεν λειτουργεί. Και το ξέραμε και εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δουλέψει. Εγώ το αντιλαμβάνομαι ως πολιτικό ζήτημα. Πιο πολύ από ότι διοικητικό ζήτημα. Δύο εκατομμύρια Ισπανοί στο εξωτερικό. Μιλάμε για 25% μείωση στην εκλογική δύναμη. Και αυτό σημαίνει τεράστιο όγκο γραφειοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλη αποτυχία τη διοίκηση. Εγώ α, ζω στο Ελσίνκι σε ένα αστυνομικό τμήμα μεγάλο κοντά. Και είναι κεντρική η γειτονιά μου. Έχουμε θεσμικά όργανα. Πώς γίνεται να χάνεται το ψηφοδέλτιο. Είναι λίγο υπερβολικό για να είναι απλά γραφειοκρατικό ζήτημα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, πιστεύω. Και το να το αναγνωρίσουμε, αναγνωρίζοντας ότι το σύστημα δεν λειτουργεί, μπορούμε να περάσουμε σε ένα καινούριο σύστημα. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει δυνατότητα να βοηθήσει. Δεν θεωρώ ότι είναι εσωτερικά αποκλειστικό το ζήτημα αποκλειστικά ιστορικό ζήτημα της Ισπανίας και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας συμβιβασμός από όλες τις πλευρές. Και αν η Ευρώπη μπορούσε να ενώσει τις δυνάμεις της θα ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης. Και πάλι σας ευχαριστώ που μου δίνετε ελπίδα. είναι το Καταρχήν, να αποστείλουμε μία επιστολή στις Ισπανικές Αρχές, όπως προελέχθη, εξηγώντας ε, τη συλλογιστική μας και ζητώντας ε, να βελτιωθεί η διαδικασία. Επίσης, όπως προελέχθη, να αποστείλουμε στην Επιτροπή Αναφορών του, της βολής των αντιπροσώπων μία επιστολή σε σχέση με το θέμα και να ζητήσουμε μία νομοθετική πρωτοβουλία από τη βολή των αντιπροσώπων. Και επίσης να ζητήσουμε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων μία γνωμοδότηση για αυτό το θέμα έτσι ώστε να καλύψει ολόκληρη την Ευρώπη. Εντάξει, ωραία, η Μπεατρίθ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις πρωτοβουλίες αυτές που θέσατε. Θα ήθελα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε επαφή με τα σχετικά Υπουργεία στα κρατημέλη και να, συμπεριλάβει και την Ισπανία κάτι το οποίο δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Ωραία. Οπότε παραμένει ανοιχτή αναφορά, έτσι δεν είναι. Ναι, λέει η Πρόεδρος, παραμένει ανοιχτή και εκκρεμούν αυτές οι τέσσερις διαδικασίες. Λοιπόν, προχωρούμε. Ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε και τους αναφέροντες. Εξετάζουμε τώρα την 1292 κάθετος 2015 εξ ονόματος του Γιώργεν Τόρμπαλ, Δανού για την απώλεια δικαιώματος ψήφου για τους Δανούς πολίτες που μετακομίζουν σε άλλη χώρα. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Και πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Παναγόπλος έχει το λόγο. Ναι. Μόνικα, perdón. Η Μόνικα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι. Η Δανία είναι από τις χώρες που δεν επιτρέπουν στους Δανούς να ψηφίζουν όταν μετακομίζουν σε άλλη χώρα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα όταν μίλησα για τους Ισπανούς αναφέροντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο δικαίωμα του εκλέγην. Πρέπει να επαναλάβουμε ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα να παρέμβουμε στην ε, ε, εθνική νομοθεσία για τις εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρέμβει ως προς την αρμοδιότητα ε, μόνο για θέματα ευρωεκλογών και τοπικών εκλογών, αλλά όχι εθνικών εκλογών. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει παράβαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος. Η Μάργαρετ, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν ξέρω που είναι οι αναφέροντες αυτή τη στιγμή, όμως το Σύνταγμα της Δανίας είναι ξεκάθαρο και αναφέρει ξεκάθαρα ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα του εκλέγην στη Δανία αν είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Πρέπει κανείς να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα εκεί όπου πληρώνει τους φόρους του. Και αυτό δεν θα αλλάξει στο Σύνταγμα της Δανίας, το οποίο δεν τροποποιείται τόσο εύκολα. Επομένως αυτό το οποίο εξετάζουμε είναι να έχει κανείς διπλή υπηκότητα. Να ε, δώσει το δανέζικο διαβατήριο και να έχει άλλη ηθαγένεια. Από ό,τι μου λένε ο αναφέρον ζει στην Ελβετία. Στην Ελβετία έχει κανείς το δικαίωμα να ψηφίσει στις ευρωεκλογές γιατί είναι δανός πολίτης Ενδεχομένως. Τίθεται αυτό το ερώτημα. Αν έμενε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να ψηφίσει στις ευρωεκλογέ. Αλλά στην Ελβετία δεν ξέρω αν παρόλο αυτά αν μπορεί να ψηφίσει στις ευρωεκλογέ. Δεν είχα χρόνο να το διερευνήσω. Ε, πάντως προτείνεται να παραμείνει ανοιχτή ή κλειστή η αναφορά. Θέλετε να τη διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά ή να την κλείσουμε. Δεν μπορούμε κάτι να κάνουμε εδώ. Είναι θέμα, πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα της Δανίας. Δεν έχει νόημα να σκέφτεται κανείς κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα να γίνει κάτι τέτοιο. Μήπως υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές τουλάχιστον, παρόλο που δεν ζει σε καμία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι τέτοιο. Θα με εξέπλητε ε, να μπορεί κανείς να συνεχίσει να ψηφίζει μέλη του το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ ζει σε χώρα που δεν είναι ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί αυτό να διευκρινιστεί παρακαλώ. Ο κύριος Πίτερ. Η κυρία Πίτερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα δεν είναι ζήτημα στο οποίο να μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω ότι δεν είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολείται με τις εκλογές της 11 Νοεμβρίου της περασμένης χρονιάς. Ψηφίσαμε ένα ψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ψηφίσαμε και για τα θέματα δικαίου. Όλα αυτά τα δικαιώματα εντάσσονται στο πεδίο των ενδιαφερόντων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Αν παραμείνει ανοιχτή δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Ούτως ή άλλως το Ευρωκοινοβούλιο ασχολείται με αυτό το θέμα, ούτως ή άλλως αναλύει αυτό το θέμα, ούτως ή άλλως η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, το εξετάζει το ζήτημα. Να παραδεχτούμε ότι είναι ένα θέμα που συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Η Μαργαρίτα παρακαλώ. Θα ήθελα να μιλήσω αγγλικά. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να έχει το δικαίωμα να ψηφίσει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν ζει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι. Ε, ε, ε αν ισχύει αυτό, τότε με εκπλήσει που έγινε δεκτή αυτή η αναφορά. Δηλαδή μένει σε χώρα που δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή μένει σε χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά κάνετε δεκτή την αναφορά του να την εξετάσετε, ε, στην οποία ζητά κάτι που έχει να κάνει με το ε, Σύνταγμα της Δανίας και που είναι αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα. Θα ήθελα να μάθω το γιατί. Η Πρόεδρος, από τις παρεμβάσεις συνάγω το συμπεράσμα ότι πρέπει να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Θα ήθελα να σημειώσω ότι εστάλει επιστολή στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας να μας εξηγηθεί αυτό που μας εξήγησε η Μάργαρετ. Επομένως, αν συμφωνείτε, δίνουμε στον αναφέροντα τις επιστολές της μόνιμης αντιπροσωπείας και τις εξηγήσεις της. Καλώς, περνούμε. Στην επόμενη αναφορά 0171-2016 του Michael Βίλιαμ Mansfield, Βρετανική Ιθαγένεια, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου των πολιτών της ΕΕ όταν είναι κάτοικοι με φορολογική κατοικία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αναφέρον δεν έχει έρθει, αλλά θα δώσουμε το λόγο και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Μόνικα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει γραπτός. Σημειώνουμε τις προτάσεις του αναφέροντος σε ό,τι αφορά ε, το δικαίωμα του εκλέγει για τους κατοίκους που ζουν σε άλλη χώρα μέλος και τη δυνατότητά τους να συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σήμερα. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο το λόγο? Καλώς. Είναι η ίδια περίπτωση με τις προηγούμενες. Κλείνει αυτή η αναφορά και περνούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ομάδα εργασίας για θέματα ευζοίας των παιδιών. Αναφορές που σχετίζονται με τις αποφάσεις της υπηρεσίας πρόνοιας για τα παιδιά και τους νέους, Jugendamt, ή και τη γερμανική δικαιοσύνη επί οικογενειακών θεμάτων. Έχουμε έκθεση της Προέδρου ε, της Ομάδας Εργασίας και στη συνέχεια θα δώσουμε λόγο σε διάφορους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Ελεονόρα Λέβη έχει το λόγο που είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που είναι εδώ παρόντες, καθώς και τις γερμανικές αρχές οι οποίες έχουν έρθει σήμερα εδώ στη συνεδρίασή μας. Το θέμα της υπηρεσίας πρόνοιας για παιδιά και νέους, Jugendamt, η υπηρεσία αυτή αποτέλεσε το αντικείμενο ε, της εργασίας μου, της εξέτασής μου διότι έχουν υποβληθεί αναφορές από διάφορους Ευρωπαίους πολίτες για το θέμα αυτό και στόχος της ομάδας εργασίας ήταν να προβεί σε μια συστημική ανάλυση για να εξετάσει το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση. Στην τελευταία συνεδρίαση της ομάδας εργασίας παρουσία των εμπειρογνωμών και των ειδικών που, είχαν που είχαμε ε, ε, προσκαλέσει για αυτό το σκοπό, ε, υπήρξε διάσταση απόψεων και θα ήθελα να σας αναφέρω αυτές τις διαφορές. Η μία ομιλήτρια μίλησε για τον πολύ διάζοντα χαρακτήρα, μοναδικό χαρακτήρα του συστήματος του γερμανικού και δεν υπάρχει αντιστοιχεία σε άλλα νομικά ειδικητικά συστήματα στην Ευρώπη. Έχουμε το δικαίωμα της πολιτοφυλακής, για παράδειγμα. Έχουμε την κυδαιμονία επί της περιουσίας και επί του προσώπου, γονική ε, Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες δηλαδή και όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν αμφιλεγόμενες διαμάχες και παραβίαση των δικαιωμάτων των ανηλίκων ή των γονέων τους, ειδικότερα όταν οι γονείς δεν είναι Γερμανοί. Από εκεί και πέρα, ειδικό έδειξε πως η σχέση μεταξύ γονιού και παιδιού αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωμης τάξης. Το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο αλλά και το δικαστήριο στο Στρασβούργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύουν αυτό το ε, δικαίωμα. Επομένω, με δεδομένο το ρόλο της υπηρεσίας πρόνοιας και την αρμοδιότητα της υπηρεσίας αυτής σε θέματα οικογενειακού δικαίου θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετίζεται με την υπόθεση. Η σχετική δικός επανήλθε στο θέμα του δικαιώματος των ανηλίκων και του δικαιώματος υπεράσπισης τους σε δίκες που γίνονται στην ε, Γερμανία ε, σε σχέση και με το δικαίωμα της, για την οικογένεια. Έρχομαι τώρα στις επικρίσεις που μας παρουσίασαν στην ομάδα εργασίας και ελπίζω οι γερμανικές αρχές να μπορούν να μας διαφωτίσουν. Ε, ποιες είναι οι αιτιάσεις δηλαδή, Πρώτον, απουσία επίσημων στατιστικών στοιχείων και λυπούμαστε γι' αυτό. Δεν υπάρχουν είτε σε ομοσπανδιακό επίπεδο είτε σε επίπεδο κρατηδίων. Δεν υπάρχουν στατιστικά που θα μας επέτρεπαν να καταλάβουμε ποια είναι η ηθαγένεια του γονιού που αποκτά την κυδαιμονία του παιδιού όταν οι γονείς είναι διαφορετικές ηθαγένειας. Γιατί τέτοια δεδομένα δεν υπάρχουν. Οι γερμανικές αρχές ε, δεν θεωρούν απαραίτητο να γίνει έρευνα για το θέμα αυτό. Καλό τις γερμανικές αρχές να μας δώσουν τα στοιχεία ε, που έχουν. Και καλό τις γερμανικές αρχές να εξετάσουν τα στοιχεία στα οποία κατέληξε η δική μας επιτροπή, η δική μας ομάδα εργασίας. Η Jugendamt, η υπηρεσία πρόνοιας, θεωρείται ότι λειτουργεί υπό την αιγίδα, υπό την αρμοδιότητα μίας διοικητικής οργάνωσης σε επίπεδο κρατηδίων. Η Jugendamt δρά επίσης και βάσει των αρμοδιοτήτων των κοινοτήτων, των δήμων. Όμως, στις συνεδριάσεις που γίνονται κάθε ε, χρόνο, πολιτική απόφαση είναι να λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικό κρατήδιο. Η Jugendamt ε, αναφέρεται στην Land Jugendamt. Πρέπει να ξέρουμε με ποιες οργανώσεις συνεργάζεται, ποιοι είναι οι υπάλληλοι της, ποιες είναι, ποιοι είναι οι φορείς που σχετίζονται με αυτήν και ποιος είναι ο προϋπολογισμός της. Θα μπορούσαμε να έχουμε στατιστικά στοιχεία και έτσι θα καταλάβουμε καλύτερα πώς είναι οι ανήλικοι ε, που εντάσσονται στην υπηρεσία αυτή κάθε χρόνο. Είναι ουσιαστικά ο τρίτος γονιός, γιατί είναι ε, διάδικο μέρος σε κάθε ε, οικογενειακή διαφορά. Αυτό προβλέπεται από τη γερμανική νομοθεσία κάθε φορά που γίνεται δικαστήριο για την κυδαιμονία των παιδιών. Ακόμα και όταν οι γονείς ασκούν όλα τα δικαιώματά τους για τα παιδιά. Και αυτό είναι ιδιαίτερο στη γερμανική νομοθεσία, δεν υπάρχει στις άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε σε ποιο σημείο της διαδικασίας η Jugendamt υποβάλλει στο δικαστή τις συστάσεις της. Ποιες είναι οι συστάσεις. Ο δικαστής, ο Γερμανός, δεν έχει επιλογή, είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις συστάσεις της υπηρεσίας πρόνοιας και τη γνωμοδότησή της. Είναι αρμόδια για την εκτέλεση επίσης των δικαστικών αποφάσεων έχει το δικαίωμα να τις ερμηνεύσει με, με, λιγό, με πιο περιοριστικό τρόπο ή με πιο ευρία ερμηνεία. Έχει αυτή τη διακριτική ευχαίρεια η υπηρεσία πρόνοιας. Ε, μερικές φορές η απόφαση παίρνει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να βγει και έτσι ε, καταστρατηγείται το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη και ε, απόφαση της δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ποιες είναι οι πρακτικές λεπτομέρειες, πότε παρεμβαίνουν οι γερμανικές αρχές, πώς παρεμβαίνουν παρεμβαίνουν για να αποφύγουν την καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η υπηρεσία πρόνοιας νομικά μπορεί να εκδώσει βουλεύματα, αποφάσεις για προσωρινά μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν την εκτέλεση μιας απόφασης του δικαστηρίου. Χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των γονιών. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά που διαφέρουν από τις άλλες χώρες και θα πρέπει οι γονείς να μπορούν να προσφύγουν εναντίον αυτών των μέτρων αμέσως. Και μερικές φορές αυτό γίνεται μετά από πολλούς μήνες, όταν ήδη έχει εδρεωθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Φάνηκε επίσης ότι οι υπηρεσίες πρόνοιας μπορούν να αξιολογήσουν τις ε, επιδόσεις των δικαστών ε, σε ό,τι αφορά το οικογενειακό δίκαιο. Δηλαδή, υπάρχει επιρροή στη σταδιοδρομία των δικαστών. Αυτό θα ήταν καλό να το γνωρίζουμε. Μιλήσαμε και για τις ακροάσεις των ανηλίκων, όταν υπάρχουν δίκες βάσει οικογενειακού δικαίου. Και είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ε, δεν ε, ηχογραφούνται οι ακροάσεις αυτές. Ούτε οι γονείς μπορεί να είναι παρόντες, ούτε οι δικηγόροι. Παίρνουν μόνο μία σύντομη περίληψη αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις. Η αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται στο εξωτερικό συστηματικά γίνεται αντικείμενο άρνησης από τις γερμανικές αρχές εάν δεν έχει υπάρξει ακρόαση του ανηλίκου, ακόμα και αν ο ανήλικος είναι εξαιρετικά μικρός, γιατί η ακρόαση είναι από τριών ετών και πάνω. Θα ήθελα να επανέλθουμε στον ορισμό και στην ερμηνεία του Kindenswall, κάτι το οποίο είναι αρκετά προβληματικό θα έλεγα με βάση ποιες αρχές δρά η υπηρεσία πρόνοιας και αν, είναι, αν δρά για την ε, ευημερία του, του ανηλίκου, πώς ορίζεται αυτή η ευημερία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωμη θα πρέπει οι δημοτικές αρχές να σεβαστούν ε, ε, όλα αυτά που προβλέπονται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ένα αίτημα άρνησης του δικαιώματος και η δαιμονίασή του δικαιώματος επικοινωνίας του γονιού θα πρέπει να ορίζεται και να εδράζεται στην ανάδειξη σαφούς κινδύνου για το παιδί και όχι με βάση ε, κάτι που αποτελεί κάτι που νομίζει κάποιος ή που είναι επεπίθεση του μόνο. Πολύ συχνά όμως υπάρχουν αμφισβητήσεις από τους αναφέροντες γιατί γίνεται λόγος για παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και των γονέων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ε, bystand. Ε, δεν γίνεται λόγος μόνο για θέμα κυδαιμονίας. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, έχει ορίσει το θέμα η γερμανική νομοθεσία σε σχέση και με τους δύο γονείς. Το Beistandschaft είναι μια διαδικασία που επιτρέπει μόνο μερός το Jugendamt να προβάλλει συγκεκριμένες πράξεις δεσμευτικού χαρακτήρα. Γι' αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε κατά πόσο οι γονείς έχουν την δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ένστασης και στην περίπτωση του ανηλίκου κατά πόσο ο γονέας ε, μη γερμανικής υπηκότητας μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Μία τελική πτυχή αφορά τις μεταφράσεις. Από όσο γνωρίζουμε, οι γερμανικές, τα γερμανικά δικαστήρια δεν ε, μεταφράζουν αυτές τις ε, κοινοποιήσει κάτι το οποίο μέσα στα πλαίσια διασυνοριακών ε, ρυθμίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι θα πρέπει να γίνεται κατανοητό το όλο θέμα και από τον κάτοικο ο οποίος δεν έχει τη γερμανική ηθαγένεια. Εάν αντιταχθεί ο παραλήπτης ζητώντας ε, τη μετάφραση, τότε τα γερμανικά δικαστήρια θεωρούν ότι θα πρέπει να αναλάβει το κόστος της μετάφρασης ο παραλήπτης. Γιατί διαφορετικά παραβιάζεται ο νόμος 1393 του 2007. Θα ήθελα λοιπόν να βοηθήσω την εργασία της ομάδας εργασίας και ολόκληρης της Επίτροπης ΠΕΤΗ. Ευχαριστούμε, Λεωνόρα. Θα δώσουμε το λόγο σε άλλα μέλη της ομάδας εργασίας που τον ζήτησαν. Η, η Χούλια Πιτέρα. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η φόβη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Jugendamt συμπεριλαμβάνονται σε διάφορες αναφορές. Αναφορές που έχουν αποσταλεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διάφορες επιστολές των βουλευτών περιλαμβάνουν διάφορα τέτοια στοιχεία. Τον Απρίλιο 2016 έγινε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μια σχετική συζήτηση για την ευημερία και την προάσπιση των συμφερόντων των παιδιών. Και καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθούν οι κοινωνικές παροχές και η φροντίδα για τα παιδιά. Το Νοέμβριο του 2011 έγινε ένα συνέδριο στο Βερολίνο το οποίο είχε αποτελέσματα και το πόρισμα ήταν ότι δεν είναι δυνατόν να μην τηρείται το ευρωπαϊκό και το εθνικό και το εθνικό δίκαιο από τις γερμανικές αρχές. Δεν διαπιστώθηκε ε, διακριτική μεταχείριση των γονιών και δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε απόδειξη διακριτικής μεταχείρισης. Τώρα, οι αναφορές για τη λειτουργία του Jugendamt και τα αιτήματα των γονέων αφορούν τα εξή ζητήματα. Πώς είναι δυνατόν να περάσουν περιορισμοί στην επίσκεψη των παιδιών από μη Γερμανούς γονείς. Και εκπρόσωποι του Jugendamt έχουν ε, προσκομίσει αποδεκτικά στοιχεία κατά των ε, γονέων σε ό,τι αφορά τις ακροάσεις τώρα στο Jugendamt. Ε, πολλά πράγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, η ευημερία του παιδιού δεν λαμβάνεται πραγματικά υπόψη. Πιο πολλοί εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη το συμφέροντα της γερμανικής κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν συστήνουμε την υποβολή ενστάσεων σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Jugendamt και προβλέπονται στον κανονισμό Βρυξέλλες 2 διάφορες τέτοιες δυνατότητες. Η μη αναγνώριση, η μη εφαρμογή των ε, δικαιωμάτων των ε, γονέων από άλλα κρατημέλη. Διαμεσολάβηση στην οικογένεια, διαμεσολάβηση και ακρόαση για την... τα συμφέροντα του παιδιού. Και επίσης ε, συχνά η απόφαση για το που θα παραμείνει το παιδί ή λαμβάνεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μόνο. Και οι μη Γερμανοί γονείς δεν έχουν πρόσβαση στα δικαστικά έγγραφα στα γερμανικά. Ουσιαστικά δηλαδή υποστηρίζονται αυτοί οι οποίοι με άδικο τρόπο ενδεχομένω μετέφεραν το παιδί στη Γερμανία. Και δεν φαίνεται ότι το Jugendamt είναι μια πολιτική, ένα πολιτικό ίδρυμα το οποίο ασκεί υπερβολικά μεγάλη πίεση. Συστάσεις τώρα για τη δραστηριοποίηση σε ό,τι αφορά την προσκόμιση τεκμηρίων για τους γονείς. Το έτος 2015 εφαρμόστηκαν μέτρα. Πριν από ένα μήνα ακούσαμε τους εμπρογνώμονες της Γαλλίας και της Ιταλίας νομομαθείς οι οποίοι τοποθετήθηκαν για τη διαδικασία σε ό,τι αφορά το Jugendamt. Και η κυρία Κολόμου επίσης κατέθεσε αναφορά την οποία στην συνέχεια απέστηρε γιατί και ότι δεν ήταν αντικειμενικός κριτής και ότι είχε ιδίων συμφέρον. Το θέμα λοιπόν αυτό το έθεσαν οι αναφέροντες. Πάρα πολλές λοιπόν είναι αναφορές από το 2015 και η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε τότε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και να αναμείνει την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέθηκε και το θέμα της αναθεώρησης και της εξέτασης του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Ο κανονισμός λοιπόν αυτός Πέρασε από τη δικασία αναθεώρησης, έγιναν διαβουλεύσεις, αμφισβητήθηκαν πολλά στοιχεία και έγιναν διάφορες έρευνες τα τελευταία πέντε χρόνια και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στράφηκε προς ε, την ε, Επιτροπή Αναφορών και τελικά προκύπτει ότι δεν υπάρχουν τεκμήρια για εμπλοκή σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Οι κεντρικές αρχές λοιπόν και οι βασικές αρχές για τη διασυνοριακή μεταφορά των παιδιών σε ό,τι αφορά μεικτά ζευγάρια. Όλα αυτά ρυθμίζονται από τη συνθήκη της Χάγης. Η Επιτροπή Αναφορών θα αποστείλει μία ένσταση. Αυτό τουλάχιστον ε, απαιτείται. Και έχω μπροστά μου την ε, ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της κυρίας Ρέντινγκ της Επιτρόπου και των αρμόδιων υπουργών, του αρμόδιου υπουργού στη Γερμανία. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να παρακολουθήσουμε επί τόπου το πώς ε, δυστυχώς ε, η ομιλήτρια διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Ζητάει συγγνώμη η ομιλήτρια decyzje, które odnoszą się do umieszczenia dziecka w instytucji niemieckiej. για την παραμονή του παιδιού στα γερμανικά θεσμικά όργανα και τα σχετικά δικαιώματα επίσκεψη δεν ρυθμίζονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προδιαγραφές τη χάρτα χάρτας βασικών δικαιωμάτων διευκρινίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο σε περίπτωση που εφαρμόζονται τα κοινοτικώς προβλεπόμενα σε εθνικό επίπεδο. Το μοναδικό δίκαιο που έχει η Επιτροπή Αναφορών είναι τα όσα αφορούν το Δικαστήριο Θεμελιντών Δικαιωμάτων σε περίπτωση που θεωρείται ότι δεν τηρείται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές των Βρυξελών 1 και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Εθνική Διαδικασίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη αποτελεί ενδικό μέσο των δικαστηρίων. Και πρέπει να γίνονται έλεγχοι και πρέπει φυσικά να διασφαλίσετε ότι υπάρχει αναλογικότητα σε περίπτωση έκδοσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Σύλληψης. Οι αναφέροντες θεωρούν ότι η γερμανική νομολογία δεν τηρεί τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α και τον κανονισμό για την αναγνώριση της νομολογίας. Καθώς και το θέμα της καταβολής διατροφής. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα ρυθμίζει το δικαστήριο του τόπου όπου ζει το παιδί. Και σε γενικέ ε, γραμμέ αυτό είναι εκεί που είναι η ζωή του παιδιού και η διαβίωση του. Η αναφορά τη λάβαμε από τη Γερμανία. Η αναγνώριση τώρα των δικαιωμάτων του γονιού, τα δικαιώματα επίσκεψης σε περίπτωση γάμου, ή σε περίπτωση έλλειψης γάμου, όλα αυτά ρυθμίζονται από τα δικαστήρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στους συντάκτες της αναφοράς να αναφερθούν στα αρμόδια δικαστήρια και να κάνουν έφεση. Και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τότε μπορεί να παρουσιαστεί η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Στρασβούργο για τα, ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α, το θέμα της νομολογίας και πώς ρυθμίζεται. Εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Όλα αυτά λοιπόν προδιαγράφονται και θα πρέπει να τηρηθούν και με συγγνώμη που μίλησα γρήγορα. Euh, Ευχαριστώ τους αναφέροντες. Ευχαριστώ και την Εύη γιατί μας μίλησε για την ε, εργασία τους. Εγώ δεν θέλω να το παίξω politically correct. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, είτε αρέσει είτε όχι. Κάναμε αυτή την εργασία γιατί εδώ και πολλά χρόνια πολλοί γονείς μη γερμανικής υπηκότητας προβαίνουν σε καταγγελίες ε, ότι δεν εισακούονται. Μιλάμε ε, και στην ουσία επιτιθέμεστα σε ε, ένα τότεμ. Πρόκειται για το Jugendamt, αυτή την υπηρεσία πρόνοιας η οποία φοβίζει. Μιλάμε Ε, μιλάμε για ευαίσθητα ζητήματα τα οποία και έτσι αντιμετωπίζονται από τις γερμανικές αρχές. Εδώ δεν καταφερόμαστε κατά της γερμανικής νομοθεσίας αλλά μιλάμε για τα δικαιώματα των γονέων και του παιδιού. Βεβαίως η ευημερία των παιδιών είναι το κερασάκι στην τούρτα πάντα. Αλλά το παιδί πρέπει να έχει το δικαίωμα να μπορέσει να ζει και να βλέπει και τους δύο γονείς. Δυστυχώς όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο με βάση και τους αναφέροντες. Οι αναφέροντες που προσέρχονται, οι οποίοι πλήττονται άμεσα, που πολλές φορές δεν έχουν ούτε νέα από τα παιδιά τους, είναι η άκρη του παγόβουνου, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν γνωρίζουν καν τα δικαιώματά τους. Και πολύ συχνά αυτό που επιβάλλει το Jugendamt είναι να αναλάβει τα έξοδα και και τη διατροφή ο γονέας ο οποίος δεν είναι Γερμανός. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά θα πρέπει να σπάσουμε αυτό το απόστημα για το Jugendamt. Μόνο οι Γερμανοί γονείς είναι καλοί γονείς, οι άλλοι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της αγάπης οι γονείς που δεν έχουν γερμανική υπηκότητα. Μιλάμε για το συμφέρον του παιδιού ή το συμφέρον του κράτους, γιατί μιλάμε και για τον τρίτο γονέα, το κράτος. Τι σημαίνει η ευημερία του παιδιού, δικαιώματα του παιδιού. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτό και μόνο αυτό. Λυπάμαι που ε, γίνομαι και ε, απότομος, αλλά Όλα τα άλλα είναι φλιναφήματα. Μας ενδιαφέρει το καλό του παιδιού. Ε, δεν υπάρχει ευημερία για το παιδί εάν του απαγορεύεται να δει έναν από τους δύο γονείς, εκτός αν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του. Αλλά εάν υπάρχει έκδηλη πρόθεση να απαγορέψουμε σε ένα παιδί να δει τον άλλο γονέα, τότε καταστρατηγούμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Ωραία. Εξόντως των Πρασίνων έχει το λόγο η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ και καταρχάς να ευχαριστήσω τους αναφέροντας. Να τους ενθαρρύνω. Και θεωρώ ότι θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση καινούργιε ευκαιρίε. Την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη Ολομέλεια, εγκρίναμε μία έκθεση τη Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ, την έκθεση Ιντφέλντ. για την ίδρυση ενός νέου σώματος, το οποίο θα εξετάζει αναχώρα το τι είναι απαραίτητο και τι ενδεχομένω θα μπορούσε να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων. Και σχεδιάστηκε λοιπόν για να ξεπεραστεί ακριβώς το πρόβλημα των διατάξεων του χάρτη των δικαιωμάτων και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Υπάρχει και πρόβλημα σε ό,τι αφορά την οριζόντια οδηγία για την ε, μη διακριτική μεταχείριση. Αν μπορούσαμε να αποτεχτούμε την ε, τις διτάξεις που αφορούν μεταξύ άλλων και άλλα πράγματα και την απασχόληση. θέματα οικογενειακά, Jugendamt κτλ. Να αναφερθώ και στην πρόταση του κυρίου Πιτέρα, της κυρία Πιτέρα, για να στραφούμε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όντω, ενδεχομένω να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά οικογενειακέ υποθέσει και τα παιδιά. Οι διαδικασίε αυτέ παίρνουν τουλάχιστον δύο χρόνια. Και ξέρετε για τα παιδιά δεν είναι αποδεκτό χρονικό διάστημα αυτό. Δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού να περιμένει μέχρι να ληφθεί η απόφαση. On behalf of one of its parents violating the... Από την απόφαση που ενδεχομένω να λαμβάνει ένα γονιό ει βάρο του άλλου. Τα λάβαμε λοιπόν αυτά υπόψη. Όσο Επιτροπή Αναφορών κρατούμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Στρεφόμαστε και προς τις αρχές. Και ξέρω ότι δεν έχει βελτιωθεί τίποτα από την διερευνητική αποστολή μας και μετά. Ίσως θα πρέπει να διοργανωθεί και άλλη διερευνητική αποστολή πριν αποφασίσουμε. Ευχαριστούμε, λέει και η Πρόεδρος. Περνάμε τώρα στους αναφέροντες πάλι θα τους ζητούσα να παρέμβουν για τρία λεπτά ο καθένα. Ε, αλλά Κυρία Ντελφίνα Παγκό, θα διαβάσει την παρέμβασή μου γιατί εγώ δεν έχω την όρασή μου. Θα ήθελα να πω ότι πέρσι χρειάστηκε να απαντήσω στις βαβαρικές αρχές, στο Jugendamt. Όμως το ε, Υπουργείο δεν δέχτηκε να απαντήσει. Τώρα έλαβα ένα γράμμα από την Επιτροπή στα Αγγλικά όπου αναφέρεται ότι δυστυχώς ε, δεν θα γίνει δεκτή η αίτησή μου. Και κάποτε αργότερα θα λάβω ένα γράμμα στα γαλλικά. Το 2012 η αίτησή μου θεωρήθηκε παραδεκτή. Σήμερα με τα τρία χρόνια μου ανακοινώνουν ότι δεν είναι παραδεκτή γιατί δεν είναι αρμόδια η Επιτροπή. Αυτό μου το ε, αναφέρει ένας Γερμανός υπήκος από το Μόναχο, εκεί που εκδικάστηκε και η υπόθεσή μου. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, είναι οι ίδιοι που χειρίστηκαν και το ζήτημα δανών υπηκών. Δυστυχώς ελέγχθη ότι αυτή η αίτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή ούτε για μας ούτε για τους δανούς. Πώς η Επιτροπή θα βρει μία λύση εάν η Γερμανία αρνηθεί να δεχτεί μία αίτηση θα ήθελα να υποβάλω στην Επιτροπή την ανταπάντησή μου προς τον κύριο Καν, ο οποίος είναι γραμματέας στη ε, Βαβερικές Αρχές Προστασίας του Καταναλωτή. Σε αυτή την ανταπάντηση έδειξα την ε, κακή θέληση του Γερμανικού Υπουργείου και μίλησα και για την ε, μεροληπτική στάση των ψυχολόγων. Αυτές οι ψευδο ψευδοπραγματογνωμοσύνες στοιχίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ και πρόκειται για μια πραγματική επιχείρηση. Η ομάδα εργασίας και η επιτροπή σας θα, θα βρουν και τα άρθρα του τύπου και τα δεδομένα του ψυχολόγου του δόκτωρα Λάιτνερ που είναι παγκοσμίως γνωστός. Ε, Λιονέλ Τζιμπέρτι 1684 του 13. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να, χαιρετήσω τα χιλιάδες θύματα του Jugendamt θα ήθελα καταρχήν να μην ε, υποβιβάσουμε το πρόβλημα που πλήττει που αφορά τη Γερμανία. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να αντιληφθούμε τους κινδύνου του οποίους εκτιθέμεθα όταν μιλάμε για τους μηχανισμούς της ε, οικογένειακή ε, δικαστικής δύναμης στην Γερμανία. Kinderklau σημαίνει ε, κλοπή των ε, παιδιών. Δεν ε, ήταν κάτι που το επινοήσαμε. Το βλέπουμε στο Google και εκατοντάδες ε, σελίδες και θα ήθελα κατευθείαν να παρακαλέσω τους διερμηνείς να μην ε, μεταφράζουν τους γερμανικούς όρους όπως Kinderklau, Jugendamt, Kindeswohl γιατί πρόκειται για πράγματα τα οποία δεν μεταφράζονται γιατί είναι συγκεκριμένα με στη δικαστική πραγματικότητα της Γερμανίας. Ε, και θεωρώ ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο διάφορες επιτροπές ε, που ασχολούνται με το θέμα αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν τις βασικές αρχές του προβλήματος. Στο 2011 υπήρξε ένα εγγραφό εργασία, το οποίο ο βουλευτής 2011 α, μας το έδειχνε και μας έλεγε ότι είχε επιληφθεί το θέμα του Jugendamt επανειλημμένα. Το Δεκέμβριο λοιπόν του 2011, τέτρες σελίδες σε ένα άρθρο του Spiegel ε, κατά το ε, ΣΕΟΥΝΤΕ σε ό,τι αφορά του γονεί που είχαν πέσει θύματα του Jugendamt. Το 2012 ο κ. Ράινερ Βίλαντ ε, προσέβαλε τον κύριο Καρέρ και τον είπε εγκληματία και τον κατηγόρησε για τρομοκρατία και συνωμοσία. Κανεί ε, βουλευτή δεν βγήκε να διαμαρτυρηθεί το 2012 επίση σε ό,τι αφορά ένα ρεπορτάζ στην γερμανική τηλεόραση με πολλές ε, με πολλά άτομα. Τον Φεβρουάριο του 2012 το δικαστήριο του Μονάχου κατηγορεί το δικαστήριο του Μιλάνου στην Eurojust και ο εισαγγελέας ο Ιταλός ε, πάει στη Χάγη για να κατηγορήσει, να προσαγάγει τις αποφάσεις του Μονούχου και ο κύριος, η κυρία Κολόμπο έφυγε από τη Γερμανία δήλωσε ε, ότι υπήρχαν προβλήματα από τον Φεβρουάριο του 2012 με τον Μάιο του 2010 και ε, αναφέρονται αναφέροντες παρακολουθούνται τηλεφωνικά στην Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και τον Απρίλιο του 2010 η κυρία Χάιντς, μια Αμερικανή που της είχαν κλέψει την κόρη, την κόρη στο Μόναχο, τη λάμβανε στην Ρώμη. Τον Ιούλιο του 2012 μετά από τις εκλογές στη Γαλλία. Ε, εκδίδονται μια σειρά ενταλμάτων από το δικαστήριο του Μονάχου κατά του κυρίου Καρέρ, του κυρίου Τζιλμπέρτη, του Δοκτρα Γικού, του κυρίου Θεωρό Χάδη, τη κύρια Καλίνα, τη κυρία Προτέκβιτς. Και τα διαμερίσματα των ατόμων αυτών τα ε, εξετάζει η αστυνομία και τους ε, απειλεί τον Ιούλιο του 2012 ο κ. Καρέ συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Ο κ. Ζιλπέρτη τον Οκτώβριο του 2012 επίσης συλλαμβάνεται και φυλακίζεται και χάνει και τη δουλειά του. Και η έφεση του κατά της ε, έκδοσης της εξετάζεται μόνο από την Αγγελικά Νούσμπεργκερ, η οποία έχει γεννηθεί στο Μόναχο το Φεβρουάριο του 2013. Ο κ. Σικού συλλαμβάνεται με ευρωπαϊκό δελμά και το δικαστήριο του Μονάχου τον καταδικάζει. Τον Ιούνιο του 2013 ο κύριος Ολυμπιέ καταδικάζεται σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης από το δικαστήριο του Μονάχου. Κυρία Καλίνα, η Γερμανίδα, η οποία είχε συλληφθεί στην Ιταλία, επιστρέφεται στη Γερμανία, εκδίδεται. Τέσσερα χρόνια λοιπόν από την κυρία Καραδίο, χρόνια για την κυρία Καλίνα, 15 μήνες για την κυρία Κολόμπο, 15 μήνες για την κυρία Πόκρεπτοβιτς, Ένα μήνας για την κυρία Ίντς, 20 μέρες για την κυρία Ζιλέ, τεράστια έξοδα για τους δικηγόρους, τα δικαστήρια και τα κρατή μέλη. Και το γεγονός ότι οι αναφορές μας δεν ελήφθησαν υπόψη σοβαρά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα κόστησε πάρα πολύ σε εμά τα θέματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι έχουμε στην κατοχή μας ένα έγγραφο το οποίο προέκυψε από το δικαστήριο του Μονάχου για την καταδίκη του ΣΥΤ σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση της συνωμοσίας. Και αυτό αφορά όλα την ασφάλεια που επικρατεί στο γερμανικό κράτος. Σας ευχαριστώ. Επόμενος αναφερον 24 24-26 του 2013. Πρέπει να είμαι λίγο πιεστική γιατί τη διερμηνία θα έχουμε μέχρι τις 12.30 και το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να τις εξετάσουμε τις αναφορές. Γι' αυτό θα είμαι πιο αυστηρή για το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Η Δελφίν, παρακαλώ. Με λένε Λούκα Πουτίν, είμαι Ιταλ... Ιταλός, πατέρας ενός παιδιού που απήχθη από τη μητέρα του, με την οποία τα είχα εκείνη την εποχή. Πήγε στο σταθμό για να πει ότι θα επισκεφθεί την οικογένειά της στην Γερμανία, υποτίθεται, και θα γύριζε μέσα σε δύο εβδομάδες. Ουσιαστικά είχε σχεδιάσει να μείνει στην Γερμανία και απήγαγε την, την κόρη μου. Από τότε που έφτασε στη Γερμανία δήλωσε ότι είναι μόνη μήν της κατοικία αυτή και η Γερμανία για εκείνη και για την κόρη μου. Η Jugendamt μου έγραψε μέσω του Job Center από το Τρεβ απαιτώντας ε, χρήματα, απαιτώντας να τους ανακοινώνω τα εισοδήματά μου και τα περιουσιακά μου στοιχεία πριν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δικαιοσύνη. σα βάζω συνημένα έγγραφα και με έκαναν τα οφειλέτη ότι δεν πληρώνω τη διατροφή, ενώ δεν υπήρξε ποτέ δικαστική απόφαση να πληρώσω διατροφή. Ούτε πριν, ούτε κατά, ούτε μετά την απαγωγή. Ήμουν και είμαι ο γονιός που έχει την κυδαιμονία. Παρόλα αυτά, το Jugendamt μέσα από το Job Center μου λέει ότι ανοίγει το Minds Staff, το οποίο δεν είναι ούτε κυδαιμονία ούτε διατροφή, από τη στιγμή που παραμένουν όλα τα δικαιώματά μου για την κόρη μου και δεν έχει ληφθεί ποτέ απόφαση δικαστική για θέματα διατροφής. Λίγες μέρες πιο μετά έλαβα την ίδια ανακοίνωση από την πόλη της Βρέμης και με την ανακοίνωση αυτή το Time επιβεβαιώνει ότι προσπορίζεται μέρος δικαιωμάτων πάνω στην κόρη μου, δηλαδή το, ε, την μέρημνα για την περιουσία της και τη διαχείριση τη μελλοντική της περιουσίας της. Καμία δικαστική απόφαση δεν βγήκε. Το Jugendheim απόσυρε από τη η μητέρα το δικαίωμα να διαχειριστεί την περιουσία της κόρης και το πήρε το ίδιο, η ίδια υπηρεσία. Και με απειλεί και θέλει με, απο... να με υποχρεώσει να αποκαλύψω την περιουσία μου σίγουρα θα ξέρει πόσα έχει να κερδίσει ε, εάν το παιδί μου μείνει στη Γερμανία. Ο δόκτωρ Κολόμπο με βοήθησε σε όλα αυτά τα εγχειρήματα και διαβήματα, η δόκτωρ Κολόμπο, και επειδή γνωρίζει πολύ καλά το, σύστημα, το σύστημα της Γερμανίας, κατάφερε να υπάρξει επαναπατρισμός της κόρης μου, παράλληλο που ε, το σύστημα ήταν εξαιρετικά ισχυρό. Και δεν υπήρχε καμία επαφή μεταξύ των δύο και υπήρχε και η μπλε κάρτα. Υπάρχει version stifed, ένα καθεστώς που είχε θεσπίσει το time, ώστε να αναγνωριστώ εγώ ως θύμα απαγωγής και να υποχρεωθούν οι γονείς να πληρώσουν. Σας στέλνω όλα τα έγγραφα, όλες τις παρατηρήσεις και σας ζητώ να μην μεταφράσετε αυτούς τους όρους γιατί δεν μπορούν να μεταφραστούν. Δεν υπάρχει νομική αντιστοιχία με ε, άλλες χώρες. Στις άλλες χώρες οι ε, τα παιδιά έχουν δύο γονείς και όχι τρεις όπως στη Γερμανία. δεν δίδεται πρόβλεψη για τη διατροφή. Αυτό είναι το βασικό μέτρο του οικογενειακού δικαίου και άρα έρεται εκ των προτέρων η αποτελεσματικότητα των δικαστικών διαδικασιών. Οι μη Γερμανοί γονεί που λαμβάνουν αυτή την ανακοίνωση δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνουν. Ο Ιταλός δικηγόρος δεν καταλαβαίνει τα γερμανικά, δεν ξέρει τι είναι Bersen Sat και συχνά δίνει τη χειρότερη συμβουλή. Πάρτε γερμανό δικηγόρο και ο Γερμανός δικηγόρος συμβουλεύει στους μη Γερμανούς γονείς να έχουν μόνιμη κατοικία στη Γερμανία και άρα να αναγνωρίσουν αρμοδιότητα στο νομικό σύστημα αυτής της χώρας, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ουσιαστικά το Jugendamt με αυτό το μέτρο διεισδύει στις ξένες δικαιοδοσίες, παίρνει μόνο του ένα δικαίωμα και καταστρατηγεί την αρχή της βάσης δικαίου, της νομικής βάσης. Η, ε, θέλω να επιβεβαιώσω αυτά που σας έγραψε η Δόκτωρ Κολόμπο, ότι δηλαδή ο κανονισμός το 2001 και ο αντίστοιχος του 2009 και ο αντίστοιχος του 2012 δίνουν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία τη δυνατότητα να εξάγει τα νομικά αποτελέσματα της δικής της δικαιοδοσίας και να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί τις ξένες αρχές για να εφαρμόσει δικές της πολιτικές αποφάσεις χωρίς να μπορούν οι ξένες ε, αρχές να αντιταχθούν σε αυτές τις αποφάσεις. Η Μπεάτα έχει τώρα το λόγο αναφορά 204 του 2015 για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Με λένε Μπεάτα Πόξε Πολ Λιτσμέγερ και ξέρετε ήρθα και το 2006 εδώ όταν υπέβαλα την αναφορά μου. Ο γιος μου τότε ήταν 7 ετών, ήταν πολύ μικρός. Και ήρθα και το 2007 στο Βερολίνο, ε, συνάντησα την αντιπροσωπεία της επιστολής των αναφορών. Ήρθα το 8, ήρθα το 12 και σήμερα είμαστε στο 2016. Ο γιος μου κάθεται δίπλα μου είναι 17 ετών και είναι πολύ πιο ψηλός από ότι εγώ. Και οφείλω να σας πω ότι τα κατάφερα. Ο αγώνας μου ενάντια στο Jugendamt και στο σύστημα των ε, οικογενειακών δικαστηρίων της Γερμανίας ε, έφερε καρπούς. Ξέρετε τι είναι αυτό το Jugendamt και οφείλω να σας πω ότι ο αγώνας μου ήταν εξαντλητικός, μου στήχησε πάρα πολλά, ήταν μέχρι τελικής πτώσεως. Στερήθηκα τους φίλους, την οικογένειά μου, πρέπει να τους ευχαριστήσω θερμά όσους με στήριξαν γιατί τελικά τους στέρισα από τα οικονομικά μέσα τα οποία μου έδωσαν για να μπορέσω να διεξάγω αυτό τον αγώνα ε, εδώ και δέκα χρόνια. Κανείς πολιτικός δεν με βοήθησε και αυτό οφείλω να το πω εδώ δημόσια. Αντιθέτως, οι Γερμανοί πολιτικοί έκαναν τα πάντα για να με παρουσιάσουν τα μέσα επικοινωνίας ως ε, μια εγκληματία. Ξέρετε, δέκα χρόνια γράφουν οι άνθρωποι αναφορέ ενάντια στο Jugendamt, στη Bundestag, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στο Amtag, στο Υπουργείο Δικαιοσύνη τη Γερμανία και πάντοτε παίρνουν την ίδια στερεοτυπική απάντηση. Ότι δηλαδή τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα, προσφύγεται εκεί. Επομένω, εμεί, οι γονεί, θεωρούμε ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα να κερδίσουμε ενάντια στην Γερμανική Υπηρεσία Πρόνοιας. Ε, υποβάλλονται οι αναφορές δεν φέρνουν καρπούς και ο αριθμός των παιδιών που κλέβουν τα γερμανικά γραφεία αυξάνεται δραστικά. Η κατάσταση για εμάς είναι πραγματικά δραματική. Ερχόμαστε εδώ, κλαίμε και η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η εμπειρία μας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μιλούμε για ηγεμονική εξουσία της Γερμανίας στο θέμα αυτό. Η Επιτροπή Αναφορών είναι η τελευταία ελπίδα για τους γονείς. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι με την πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχουμε καταφέρει. Απευθύνομαι λοιπόν σε εσάς, στους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητώ να κάνετε κάτι για τους Ευρωπαίους λαούς για τους Ευρωπαίους πολίτες που σας έχουν εκλέξει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να δράσετε γιατί καταστρατηγούνται ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού από την υπηρεσία πρόνοιας. Έχουμε το άρθρο 237 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και άλλα εργαλεία, έχουμε άλλα μέσα στη διάθεσή μας. Υπάρχουν όλα αυτά. Και χάρη σε αυτά τα εργαλεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει Έχουμε το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά σας συγκετεύω. απευθύνω έκκληση δραματική. Ας μην μιλούμε άλλο, ας περάσουμε στη δράση. Ευχαριστώ. Επόμενη αναφορά 437 του 2016. Ο αναφέρον έχει το λόγο παρακαλώ. Δεν είναι παρόν. Ναι, εγώ είμαι και θα διαβάσω την αναφορά του. Παρέμβαση για την αναφορά του κυρίου Γομπέρνο Τιτσιόλη. Με την αναφορά αυτή θέλουμε να, υποβάλουμε, να θέσουμε υπόψη των ευρωπαϊκών δεσμικών οργάνων το μη σεβασμό και τη μη τήρηση με συστηματικό τρόπο από τα δικαστικά και αυστριακά ε, δικαστήρια του κανονισμού 1393 του 2007 Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σε ό,τι έχει να κάνει με την γνωστοποίηση, κοινοποίηση δικαστικών και εξοδικαστικών αποφάσεων αστικού ή εμπορικού δικαίου. Τα αυστριακά και γερμανικά δικαστήρια υποχρεούνται να κοινοποιήσουν αυτή την απόφαση σε μία... Συγγνώμη, πολύ αργά λέει, κάπως πιο αργά διαβάστε αν γίνεται, λέει η Πρόεδρος, για να σας παρακολουθεί η διερμηνία που δεν έχει το κείμενο. Ε, επομένως, συνεχίζει η ομιλήτρια. Τα γερμανικά και αυστριακά δικαστήρια καλούνται να γνωστοποιήσουν τις αποφάσεις τους σε μία γλώσσα η οποία γίνεται αντιληπτή από τον παραλήπτη, από τον αποδέκτη ή στην επίσημη γλώσσα του κράτους που αιτείται την κοινοποίηση ή γνωστοποίηση. Αντιθέτως, τα ευστριακά και γερμανικά δικαστήρια γνωστοποιούν τις αποφάσεις τους στα γερμανικά στον αποδέκτη ή παραλήπτη, παρόλο που ε, ο αποδέκτης μπορεί να μην είναι γερμανός ή να μην γνωρίζει τη γερμανική γερμανικά και αυστριακά δικαστήρια μεταφράζουν τις αποφάσεις τους πριν τις γνωστοποιήσουν ή πριν τις κοινοποιήσουν. Στη συνέχεια αποστέλουν άλλη κοινοποίηση ή γνωστοποίηση καταδικάζοντας τον παραλήπτη και αποδέκτη να καταβάλει τις δαπάνες για τη μετάφραση ουσιαστικά. Και προκύπτει το εξή. Τα αυστριακά και γερμανικά δικαστήρια γνωστοποιούν την απόφασή τους στα γερμανικά στους ξένους αποδέκτες, π.χ. Ιταλούς, ο Ιταλός πολίτης αρνείται την κοινοποίηση, γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 1393 του 2007 γιατί η εν λόγω γνωστοποίηση κοινοποίηση δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε γλώσσα καταληπτή από τον αποδέκτη ή στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους που αιτείται την ε, ε, γνωστοποίηση ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης. Τα γερμανικά και αυστριακά δικαστήρια επομένως με μεταφράζουν την απόφαση του στα Ιταλικά και στη συνέχεια ε, στέλνουν γνωστοποίηση στον αποδέκτη καταδικάζοντας τον να καταβάλει την έξοδα της μετάφρασης. Ή, επίσης, τα γερμανικά και αυστριακά δικαστήρια μεταφράζουν άμεσα τις αποφάσεις του στα Ιταλικά και στη συνέχεια αποστέλνουν μια κοινοποίηση, το συνήθως στα γερμανικά, ε, στον αποδέκτη όπου τον καταδικάζουν να ε, καταβάλει τα έξοδα ναι, της μετάφρασης. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά αποτελούν σοβαρή μη εκπλήρωση, μη τήρηση του κανονισμού 1393 του 2007 από πλευράς γερμανικών και αυστριακών δικαστηρίων. Καλώς λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει η Ντελφίν Πάγο. Εκπρόσωπος της, ε, για την αναφορά 459 ε, του 2016 από τη σχετική ε, Ομοσπονδία. Καλημέρα, είμαι η Ντελφίν Πάγκο, μέλος ενός συλλόγου εξ ονόματος του οποίου παρεμβαίνω εδώ σήμερα. Ο Σύλλογος αυτός επιθυμεί να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή του Αναφορών ότι από τότε που υπέβαλε την αναφορά έμαθε και για άλλες υποθέσεις όπου οι γονείς έχουν απειληθεί και έχουν παρενόχληθεί αναλόγως. Σήμερα, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, θα εκθέσουμε εν συντομία δύο υποθέσεις που καταδεικνύουν του, λόγου του αληθές, αυτό που περιγράφουμε στην αναφορά μας. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για την κυρία Βαλέρη Σουμπισεσκή. Είναι μια μητέρα η οποία παρανόμως είδε το δικαίωμα της κυδαιμονίας να της αφαιρείται στη Γερμανία και στερήθηκε επαφή με τα δύο της παιδιά, κάθε επαφή και επικοινωνία από το 2004. Και ξαφνικά πρόσφατα καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Μπάντεν Μπάντεν να πληρώσει 6.904 ευρώ ως ληξιπρόθεσμη διατροφή και να ε, καταβάλει κάθε μήνα 348 ευρώ ανά ε, παιδί, δηλαδή 690 ευρώ περίπου το μήνα για τα δύο παιδιά. Φαίνεται η καταδίκη αυτή φαινομενικά νόμιμη και είναι απατηλή, είναι εξαπάτηση για τους κάτω θυλόγους. Πρώτον, Καταρχάς υπήρξε καταστρατήγηση παράβαση του κανονισμού 1393 του 2007, ε, κανονισμού που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 13 Νοεμβρίου του 2007, σε ό,τι έχει να κάνει με τη γνωστοποίηση και κοινοποίηση νομικών, δικαστικών και έξοδικαστικών αποφάσεων σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Πράγματι, η κυρία Τσιμπισέσκη έλαβε επιστολή από το γερμανικό δικαστήριο στα γερμανικά, μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει. Δεύτερον, έχοντα ζητήσει μετάφραση σύμφωνα με τον κανονισμό που έχει αναφερθεί, της εστάλει επιστολή μετάφρασης μαζί με το τιμολόγιο του δικαστηρίου για τα έξοδα της μετάφρασης. Τρίτον, με την ελόγω επιστολή η οποία ήταν μερικώς μεταφρασμένη και άσχημα μεταφρασμένη, το δικαστήριο τη ζητούσε να του ανακοινώσει τους οικονομικούς της πόρους μέσα σε τρεις εβδομάδες, το σύνολό τους. Τέταρτον, με την επιστολή αυτή έλαβε η λόγω και μια άλλη επιστολή του δικαστηρίου που είχε στείλει το ίδιο δικαστήριο την ίδια ημέρα που την κατηγορεί να μην τηρεί, ότι δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα και ότι αρνείται να συνεργαστεί. Και με αυτή τη βάση τη ζητήθηκε να πληρώσει πολύ σημαντικά ποσά που ε, ε ανοίγουν στη σφαίρα της φαντασίας. Πέμπτον και τέλος, κατ' εφαρμογή του κανονισμού 4 του 2009, ο πρώην σύζυγος της κυρίας Σιμπισέσκη βασίστηκε σε αυτή την ε, παράνομη απόφαση για να προσφύγει σε δικαστικό κλητήρα. Και αν δεν ήταν προσεκτική αυτή η κυρία δεν θα μπορούσε να το είχε αποδείξει ε, Δηλαδή διαβάζοντας τις δύο αυτές επιστολές θα μπορούσε κανείς να συνάγει ότι αρνείται να πληρώσει διατροφή, που ήταν θεμητό να τη ζητηθεί διατροφή, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και μία άλλη υπόθεση θέλω να σας ε, αναφέρω για ένα άτομο που έχει σταθερό εισόδημα και όπως κάθε γονιός που υποβάλλει έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυσκολεύεται ιδιαιτέρως να έχει δικαίωμα επικοινωνίας με τα παιδιά του. Η υπηρεσία πρόνοιας του ζητούσε να έχει ε, διατροφή να πληρώνει που, είναι, να ξεπερνάει τους οικονομικούς του πόρους, διότι διευκρινίζει η υπηρεσία πρόνοιας ότι τα πτυχία του και τα διπλώματά του του επιτρέπουν να κερδίσει περισσότερα χρήματα και γι' αυτό πρέπει να καταβάλει ψηλότερη διατροφή, περισσότερη από όσα χρήματα έβγαζε εκείνη τη στιγμή. Η Πρόεδρος, παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Βλέπετε λοιπόν ότι σας παραθέτουμε δύο υποθέσεις για τις οποίες οι γερμανικές υπηρεσίες ε, παίρνουν αποφάσεις με βάση απαράδεκτες αρχές από τα άλλα κράτη-μέλη και εφαρμόζονται οι αποφάσεις αυτές στο σύνολο της Ευρωπαϊκής επικράτειας για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της γερμανικής κοινότητας. Ευχαριστώ. Τέλος, εξετάζουμε την αναφορά 1021 του 2016. Παρακαλώ. Τρία λεπτά έχετε. Καλημέρα σας. Είμαι η Καρίνα Μπάσελη. Είμαι η μητέρα ε, μιας, ε, ενός κοριτσιού 12 ετών. Ο πατέρας είναι Γερμανός, δεν μπορεί να μιλήσει γαλλικά και ε, έλαβα επιστολές από το Jugendamt γιατί πρέπει να έρθω σε επαφή μαζί τους. Θέλουν να αλλάξουν ε, την ταυτότητα του παιδιού μου. Ο αδελφός της είναι εννέα ε, ετών, ζει μαζί μου στη Γαλλία και θέλουν να της αποδώσουν το νέο επώνυμο της, το επώνυμο της νέας συζύγου του πατέρα. Ε, είπα στις αρχές πώς έχουν τα πράγματα στη Γαλλία και είδα ότι κάτι τέτοιο αντιτίθεται όχι μόνο στο γαλλικό νόμο, αλλά και του νόμου γενικότερα. Εγώ έχω ένα κορίτσι 12 ετών και μπορεί να αλλάξει ταυτότητά της ε, γιατί το επιτρέπει γερμανικός νόμος. Ε, μου είπαν ότι από το προξενείο ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να θεωρηθεί προ προγονή, αλλά αλλάζει σχέση ε, μητέρας και παιδιού, βιολογικής μητέρας. Εγώ δεν είμαι φέρουσα μητέρα. Εγώ έλαβα επίσης μία επιστολή από το δικαστήριο ε, μου απεστάλλει μία ε, καταγγελία πρόσφυγη πριν λάβω το γράμμα του Jugendamt, σαν να είναι η ίδια η ενάγουσα, η ίδια η κόρη μου. Και μετά το δικαστήριο μου μίλησε για τον... Εκτός από το δικηγόρο ότι υπάρχει ένας φερφάρερ bystandum. Υπάρχει μια διαδικασία φερφάρε bystandum, την οποία δεν κατανοώ εγώ. Ε, ε, στην περίπτωση του Φερφάρεν Bystand μου λένε ότι πρόκειται για δικηγόρο του παιδιού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στα 12 χρόνια γιατί ε, όπως ξέρετε την κυδαιμονία την συμμεριζόμαστε ο πατέρας και εγώ με απασχολεί αυτή η διαδικασία και τώρα περιμένω τη συνέχεια που θα δοθεί. ως προς την κάλυψη των ε, δικαστικών εξόδων, την ε, δικαστική αρρωγή που ζήτησα, ε, μου ζητούν για κάτι τέτοιο μία μετάφραση. Θα απαντήσω στο δικαστήριο ότι εκείνοι θα πρέπει να καταβάλουν το έξοδα της μετάφρασης. Ωραία γιατί άμα υπάρχει αίτημα δικαστικής παινίας πάει να πει ότι δεν έχω τα χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ τους αναφέροντες. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στις γερμανικές αρχές. Το Jugendamt από το Βερολίνο. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η απάντησή σας σε όλες αυτές τις αναφορές. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ και κυρίε βουλευτέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν είναι απλό προφανώ. Ε, να βρίσκουμε εδώ γιατί είναι πολλαπλές οι κατηγορίες που μας έχουν απευθυνθεί και πώς να απαντήσω σε όλες τους. Θα ήθελα να παρουσιάσω το ποιος είμαι. Εργάζομαι σε ένα Jugendamt. Δεν είμαι το γερμανικό Jugendamt. Ε, εργάζομαι σε ένα από τα 12 Jugendamt του Βερολίνου. Βλέπετε λοιπόν στο χάρτη, είναι στα α, βυτικά της α, ε, πόλης. Έχουμε 170 διαφορετικές εθνικότητες και 300.000 κατοίκους εδώ. Έχουμε περίπου 130, 130 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε επίσης ε, 130 υπαλλήλου. Ε, Εργάζομαι εδώ και 20 χρόνια στο Jugendamt και πάντα υπάρχουν αμφιλεγόμενε περιπτώσεις και υποθέσει ε, και για, για πολλά χρόνια ήμουν και αναπληρωτής Γενικό Γραμματέα. Να μιλήσω λίγο για την ε, δομή των Jugendamt στη Γερμανία. Σε τρία επίπεδα βασιζόμαστε. Καταρχάς, υπάρχει το ομοσπονδιακό δίκαιο, ο κοινωνικός κώδικας υπαριθμών 8 και η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι θέμα των 16 κρατηδίων της Γερμανίας, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο. Τα Jugendamt ε, ρυθμίζονται λοιπόν ε, σε επίπεδο κρατηδίων. Περίπου 600 υπάρχουν λοιπόν τέτοια γραφεία πρόνοιας με διαφορετικό μέγεθος. Δεν θέλω να σα κουράσω με λεπτομέρειες, ε, γιατί τα πράγματα είναι και πάρα πολύ περίπλοκα σε ό,τι αφορά τη δομή των Jugendamt. Αυτό που ήταν σημαντικό είναι να διευκρινίσουμε ότι τα τοπικά κοινοβούλια ασχολούνται εντατικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία των Jugendamt και μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν και να δίνουν εντολές στα Jugendamt. Ο νόμος τώρα σε ό,τι αφορά τα Jugendamt αφορά κυρίως ε, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ε, των γονέων, των παιδιών και των νέων, θέματα εργασίας των νέων, ε, θέματα κατάρτισης, εκπαίδευση, ανάπτυξης των παιδιών κτλ. Και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ρυθμίζονται σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες εκτίκασης υποθέσεων για παιδιά. Και σκοπό είναι να υποστηρίξει την οικογένεια και του νέου ε, του Jugendamt. Στην παράγραφο 1 βλέπετε ε, τις προγραμματικές, ε, το πρόγραμμα και την ε, ερμηνεία του νόμου του άρθρου 1 του κοινωνικού κώδικα. Καθορίζει το δικαίωμα των παιδιών και των νέων για ανάπτυξη, κατάρτιση και το καθεξής. Και το βασικό είναι ότι στο επίκεντρο είναι τα συμφέροντα του παιδιού, η ευημερία του παιδιού. Είναι το βασικό σημείο προσανατολισμού για τη δράση του κράτους σε ό,τι αφορά περιπτώσεις αμέλειας των παιδιών. Ετέθησε το 2008, ρυθμίστηκε το θέμα της ε, αμέληση, αμέλειας των παιδιών. Αν, την, αν αποφασιστεί ότι υπάρχει θέμα κινδύνου για το παιδί προβλέπονται υποχρεωτικές διαδικασίες και το βασικό δικαίωμα επιμέλειας και κυδαιμονίας των παιδιών καθορίζεται από το Σύνταγμα. Δεν έχει δικαίωμα παρέμβαση στο Jugendamt στο δικαίωμα αυτό. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να ληφθούν μόνο από δικαστήριο για την παρέμβαση στην επιμέλεια. Μόνο μία εξαίρεση προβλέπεται. Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, τότε το παιδί μπορεί να δεθεί υπό επιμελητία. Αλλά θα πρέπει να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την απόφαση πάντα και ένα δικαστήριο για οικογενειακά ζητήματα. Αυτό ορίζεται και στον αστικό κώδικα, παράγραφος 50. Αλλά και εδώ δεν θα ήθελα να υπησέλθω σε λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα Τη συμμετοχή του Jugendamt ορίζεται στην παράγραφο 50, όπως σας είπα, στις δικαστικές δικασίες και σκοπός είναι η βοήθεια, η αρρωγή προς το δικαστήριο σε περίπτωση χωρισμού των γονέων και πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές συνθήκες που επικρατούν στην οικογένεια προκειμένου να βρεθεί μια αποδεκτή λύση και από τα δύο μέρη για το μέλλον του παιδιού. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν από αυτό, το βασικό είναι η ευημερία του παιδιού και όχι τα συμφέροντα των γονέων. Το οικογενειακό δικαστήριο υποχρεούται να ακροαστεί το Jugendamt. Δεν είναι υποχρεωμένο ωστόσο να ακολουθήσει τις συστάσεις του Jugendamt και οι δύο πλευρές είναι ανεξάρτητες σημαίνει από τις δε. Και ανεξάρτητα λαμβάνουν και τις αποφάσεις τους. Άρα ως εκ τούτου δεν υπάρχουν κοινέ ρυθμίσεις, συμφωνίες, επιρροές προς αλλήλους. Σε ό,τι αφορά την κυδαιμονία, οκτώ ζητήματα πρέπει να διευκρινιστούν μεταξύ των γονέων. Καταρχάς, που παραμονεμένη επίσκεψη, ε, φροντίδα, θρησκεία, σχολείο κ.ο.κ. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν ενδεχομένω είναι αμφιλεγόμενα και σε κάποιες περιπτώσεις το θέμα της υγείας, για παράδειγμα, είναι συχνά ένα σημείο για το οποίο οι γονείς πολλές φορές, ακόμα και αν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για άλλα θέματα, διαφωνούν. Η λύση λοιπόν για τις περιπτώσεις αυτές προϋποθέτει ε, διάθεση επικοινωνίας και συμβιβασμού και από τις δύο πλευρές και την ε, ανοχή και την παραδοχή σύνδεσης με τον άλλο γονέα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός κα, κανενός γονιού. Αυτό δεν προβλέπεται από τις προδιαγραφές και από τις διατάξεις. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, περίπου στο 80% καταφέρνουν οι γονείς να καταλήξουν σε μία συμφωνία σε 15-16% των περιπτώσεων μετά από ειδική αραγή οι γονείς καταλήγουν σε συμφωνία το... για τα βασικά αυτά θέματα και υπάρχουν και μια χούφτα προβληματικών υποθέσεων οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις παίρνουν χρόνια και χρόνια και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια λογική αποδεκτή λύση. Στις αμφιλεγόμενες λοιπόν αυτές τις υποθέσεις εμείς είμαστε διαμεσολαβητές από το κέντρο του Jugendamt με ψυχολόγους, με θεραπευτές όπου προσπαθούμε από κοινού με τους γονιούς να καταλήξουμε σε μια αποδεκτή λύση. Το οικογενειακό δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εφαρμογή διαφορών ε, λύσεων όπως η εξωτερική διαμεσολάβηση, αρρωγή, δικαστική αρρωγή κτλ σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις γίνεται και γνωμοδότηση των, από τους εμπειρογνώμονες. Αυτές οι διάφορες μορφές λοιπόν τώρα ως σκοπό έχουν να ερευνηθεί η ευημερία του παιδιού και το βέλτιστο αποτέλεσμα για το παιδί. Το Οικογενειακό Δικαστήριο θέλει να σχηματίσει μια σωστή άποψη για την ευημερία του παιδιού και η νομική αρρωγή δίδεται μετά από εντολή του παιδιού. Μπορούν να τα ζητήσουν και οι γονείς αυτό, δηλαδή εθελοντικά αυτό. Τα παιδιά και οι νέοι περνούν από ακρόαση, αλλά δεν υπάρχει καταγραφή, όπως σας ε, είπα, ε, των ε, ακροάσεων αυτών. Η υποχρέωση για να βρεθεί μια σενετική λύση έχει και τα όρια τη όταν διακυβεύεται η ευημερία του παιδιού, όταν τίθεται θέμα για παράδειγμα βίας, όταν δεν καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Ή υπερισχύουν ενδεχομένω το συμφέρον του κουνιού. Σε ό,τι αφορά τις εφέσεις ε, και τις ενστάσεις, υπάρχουν εξοδικαστικές λύσεις διοικητικά που μπορούν να κατευθούν στις ε, κυβερνητικές επιτροπές στο Υπουργείο Ιστορικών. Εκεί όμως δεν ελέγχεται το περιεχόμενο, ελέγχεται μόνο η διαδικασία. Αν υπάρχουν ε, ε, ενστάσεις και καταγγελίες για τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου υπαλλήλου μπορούν πάντα να υποβληθούν αυτές οι καταγγελίες σε περίπτωση σφάλματος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πραγματικά το σφάλμα αυτό, υπάρχουν διοικητικές χειρώσεις ασφαλώς. Η απόφαση του, δικαστικού, του οικογενικού δικαστηρίου μπορεί να ε, εξεταστεί επίση από τα ειδικά δικαστήρια. Και χθε από την Διεθνή Κοινωνική Επιτροπή για το θέμα των συγκρούσεων, για τα θέματα κινδαιμονίας παιδιών, έλαβα κάποια αριθμητικά στοιχεία. Μέχρι τον Οκτώβριο φέτος είχαμε 699 αιτήσει τηλεφωνικές και 56% αφορούσε απαγωγές παιδιών 29% θέματα κοινωνίας, 14% για θέματα επίσκεψης και 1% θέματα διαμεσολάβησης. Τα πιο συχνά κράτη είναι κατά 30% η Τουρκία και η ΙΠΑ, 48% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία, οι πιο συχνές χώρες και έχουμε και την Ρωσία, το Μαρόκο και την Τινησία. Είναι κάποιο συχνές χώρε Το θέμα της απαγωγής των παιδιών έχει να κάνει με τον φόβο απαγωγής. Φοβάμαι δηλαδή ότι θα μου απαγάγουν το παιδί και θα το πάνε στο εξωτερικό ή για θέματα επιστροφής του παιδιού από το εξωτερικό. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι πρόκειται για αμφίδρομα προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα κοιτάξουμε μόνο από τη μία πλευρά. Πρόκειται για προβληματικές περιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δύο υποθέσεις και αποτυπώνουν ε, ουσιαστικά διαφωνίες και φιλονικίες μεταξύ των γονέων, όχι μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Σε διάφορες περιορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ε, διαμάχες ε, πάρα πολύ οξύες το Jugendamt σε διάφορες περίπτωσεις κατηγορείται, το οικογενειακό δικαστήριο κατηγορείται, αλλά αν ε, οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την αντιμετώπιση του παιδιού, σε διάφορες περιπτώσεις δίνονται τελεσίγραφες αποφάσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των παιδιών. Σε περίπτωση διαπολιτισμικών τέτοιων συνεννοήσεων, αυτές οι πιθανότητες παρανόησης είναι ακόμα μεγαλύτερες και αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι γονείς, οποιαδήποτε λύση και να επιβληθεί απ' έξω δεν θα ικανοποιήσει κανέναν. Αυτή είναι η ουσία του θέματος και αυτό ισχύει για όλες τις γερμανικές υποθέσεις όπως και για σε όλες τις διαπολιτισμικές περιπτώσεις. Βλέπουμε ότι ο γονέας ο οποίος δεν ε, ικανοποιείται επιδεικνύει δυσαρέσκεια και κατηγορεί όλα τα θεσμικά όργανα στη συνέχεια η ε, συστηματική διακριτική μεταχείριση κάποια ομάδα γονέων είναι κάτι το οποίο αρνούμαστε κατηγορηματικά. Εγώ ποτέ δεν το έχω ζήσει προσωπικά. Αλλά φυσικά κατανοώ ότι το πολυσύνθετο της γερμανικής διαδικασίας, το γλωσσικό θέμα, τα ταξίδια, διαφορετικές νομικές πραγματικότητες μεταξύ των χωρών και φυσικά και διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις αποτελούν βάση για παρανόηση, σύγχυση και ενδεχομένω να ερμηνεύονται ω διακριτική μεταχείριση. Αντικειμενικά όμω δεν στέκει κάτι τέτοιο. Οι περιπτώσει ε, ε, διαφωνία και τη κυντεμονία παίρνουν χρόνια και περνάνε από διάφορα επίπεδα έφεση, δικαστηρία κτλ. Και πίσω από αυτό κρύβονται φυσικά τραγικέ υποθέσει, στι οποίε εμεί ω Jugendamt συχνά κάνουμε το λιγότερο εσφαλμένο, αν θέλετε. Δηλαδή, επιλέγουμε τη λιγότερο εσφαλμένη ε, δυνατότητα η έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη διαλεκτικότητας οδηγούν σε αδιέξοδα. Και η άρνηση ε, επαφής με τον ε, γονιό, με τον γονιό λόγω του φόβου απαγωγή ε, δεν επιτρέπεται να συμβαίνει. Αλλά πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα το πρόβλημα της απαγωγής και αυτό το καταδεικνύουν τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία μόλις σας ανέφερα. να σας πω και το εξής. Μπορεί μία μητέρα να κλιμακώσει την κατάσταση αρνούμενη την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα και ο πατέρας να πολεμήσει για τα παιδιά του, να στέλνει επιστολές, να στέλνει δώρα, να στέλνει email, να περιμένει το παιδί στο προαύλιο και να κάνει επιχρόνια αγώνα δικαστικό. Η μητέρα σε αυτή την περίπτωση ε, έχει παραβιάσει τα δικαιώματά της. Γιατί δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά της εναντίον της κυδαιμονίας. Αλλά τα παιδιά, για παράδειγμα, αν τα πηγαίνουν καλά κοινωνικά, έχουν φίλους κτλ. Η συμπεριφορά του πατέρα εναντίον του παιδιού ενισχύει την πίστη του παιδιού στη μητέρα και τελικά οδηγεί στην απόλυτη άρνηση και απόρριψη του πατέρα από το παιδί. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, τραγικές. Αλλά αν παίρνουμε τα παιδιά στα σοβαρά, πρέπει να λάβουμε σοβαρά και την επιθυμία τους να δουν ή να μην δουν κάποια γονέα. Η μοναδική λύση θα ήταν να βάλουμε το παιδί σε ένα ίδρυμα για να υπάρχει μια ουδέτερη, αν θέλετε, δυνατότητα επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα. Αλλά και αυτή η παρέμβαση δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται. Στην πράξη δεν επρόκειτο να το κάνουμε αυτό. Και έτσι μεταξύ των δύο αυτών γονέων συχνά ε, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αλληλοκατηγοριών και αυτό από κάποιον εξωτερικό παράγοντα δεν μπορεί να επηρεαστεί. Κατηγορία ο πατέρας, τη μητέρα, ότι δεν του αφήνει να δει το παιδί, η μητέρα ε, θεωρεί ότι από τη συμπεριφορά του πατέρα και αυτή η κλιμάκωση σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να αλλάξει. Και εδώ το θέμα δεν είναι η εθνικότητα, η υπηκότητα των γονέων. Σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεαστούν απ' έξω, επαναλαμβάνω. Το θέμα αυτό το συζήτησα πρόσφατα με δικαστές από οικογενειακά δικαστήρια και πιστεύω ότι είναι σημαντικό στο σημείο αυτό. Φυσικά αυτά είναι προβλήματα και το θέμα της διαπολιτισμικής ε, αρμοδιότητας ε, είναι σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μετεκπαίδευση και των δικαστών για να διευκρινίζονται τέτοια ζητήματα και καλό θα ήταν να υπάρχει και διεθνής ανταλλαγή των ειδικών δικαστών. Γιατί οι νομικές και οι διοικητικές οργανώσεις ε, είναι πολύ διαφορετικές σε κάθε κράτος μέλος και φυσικά δεν είναι και πολύ γνωστές ε, μεταξύ των κρατών μελών. Και να ξεκινήσουμε από το πολύ απλό, το πώς ερμηνεύεται σε κάθε χώρα το θέμα της ευημερίας των παιδιών τι δυνατότητε υποστήριξη υπάρχουν. Αυτό θα ήταν ένα ε, επικοδομητικό τρόπο να προχωρήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Θα δώσουμε... Θα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους Κομισιόν, καταρχήν από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. υπήρξαν πολλές αναφορές κατά του Jugendamt τα τελευταία χρόνια και μερικές από αυτές έχουν κλείσει και στείλαμε ε, απαντήσεις πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ακόμα στον κατάλογο. Είχαμε και μία περίπτωση πέρσι το Μάιο που αφορά ενήλικες Εάν μιλάμε για την ευημερία των παιδιών, αναρωτιέμαι γιατί μιλάμε για περιπτώσεις που αφορούν ενήλικες. Αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολες. Ποτέ δεν κερδίζει κανείς. Η Επιτροπή ελέγχει διεξοδικά κάθε αναφορά. Δεν υπάρχει μια γενικευμένη λύση και κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά. Το κύριο μέλημά μας είναι το συμφέρον, το πρωταρχικό συμφέρον του παιδιού, όπως ορίζεται και από τη συνθήκη. Χωρίς να θέλω να προδικάσω ορισμένες νέες αναφορές που δεν έχουν εξεταστεί καμία περίπτωση δεν δείχνει ότι παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο. Όπως είπα και πέρσι, μετά την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της τότε Επιτρόπου Ρέντινγκ και του Υπουργού Σρέντερ θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να γίνει ε, έρευνα σε επίπεδο Jugendamt. Θα πρέπει να το δούμε υπό την ευρύτερη έννοια στα πλαίσια της κυδαιμονίας ή της επιμέλειας του παιδιού. Βλέπουμε δυσκολίες σε πολλές χώρες και θα πρέπει να υπάρχει προστασία του παιδιού από επαγγελματικές ομάδες, από επαγγελματίες. Ίσως ε, οι μικρότερες κοινότητες ή οι δήμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να δούμε και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλαμβάνουν επαγγελματίες τα παιδιά να έχουμε μία δικαιοσύνη που να είναι φιλική προς το παιδί, όπως ορίζει και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και να υπάρχει δικαιοσύνη, απόδοση δικαιοσύνης προς το παιδί, να μην υπάρχουν ε, όρια ηλικία τα οποία να είναι αυθαίρετα και να υπάρχει προτεραιότητα περιπτώσεων, των περιπτώσεων που αφορούν παιδιά. Πολλές φορές ε, περνάνε πολλά χρόνια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν να δοθούν καλύτερες προτεραιότητες. Η Επιτροπή, όπως είπαμε και πέρσι, θεωρεί ότι ορισμένες αναφορές βρίσκονται στη δικαιοδοτική ε, διαδικασία και γι' αυτό είναι μονομερής ε, η παρουσίαση. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, τον να... κατά πόσο με το να κρατάμε αυτές τις αναφορές στην ουσία δίνουμε ελπίδες στο γονέα που έχει στην ουσία χάσει. Θα δώσω στη συνέχεια το λόγο στους δύο συναδέλφους. Να πω δύο λόγια για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2, ο οποίο αναφέρθηκε σήμερα ως ένα από τα βασικά εργαλεία που θίγονται και στις αναφορές πέρα από τα θέματα. Στο παρελθόν, λοιπόν, είχαμε συζητήσει το εργαλείο αυτό της δικαστικής συνεργασίας και κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ερευνήσει τις περιπτώσεις αυτές και να περιοριστεί μόνο σε θέματα νομολογίας, δικαιοδοσίας, αναγνώρισης, εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων χωρίς να επαναλάβω αυτά που έχουμε πει στο παρελθόν. Θα ήθελα απλά να διευκρινίσω το εξή. Η μεταρρύθμιση, η αναθεώρηση του Βρυξέλλες 2 είναι σε διαδικασία, είναι και κάποια από τα προβλήματα τα οποία αναφέραν οι αναφέροντες και οι βουλευτές περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση αυτή. Για παράδειγμα, η ακρόαση του παιδιού αποτελεί ένα από τα θέματα τα οποία εξετάζουμε στην ε, έκδοση του κανονισμού. Προκειμένου στο μέλλον να μην υπάρχουν περιπτώσεις μη αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων σε ό,τι αφορά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών για την, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές για την ακρόαση των παιδιών και επίσης η διάρκεια της διαδικασία στο μέλλον Δεν θα πρέπει οι διαδικασίε αυτέ να παίρνουν πάρα πολύ χρόνο, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι είναι προ το συμφέρον του παιδιού να είναι γρήγορε και αποτελεσματικέ αυτέ οι διαδικασίε. Και όπως είπε ο συνάδελφος, ε, δεν μπορούμε να έχουμε μία λύση για όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν και από τους ε, αναφέροντες. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνούμε. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτές οι υποθέσεις θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, μία προς μία, με την δέουσα προσοχή κάθε φορά, προκειμένου για κάθε αναφορά να υπάρχει μία συγκεκριμένη καθοδήγηση. Να διευκρινίζουμε προ τον αναφέροντα σε κάθε περίπτωση ποια είναι η καλύτερη πορεία που πρέπει να ακολουθήσει και σε ποιον πρέπει να στραφεί. Δεν υπάρχει ωστόσο μία λύση εφάπαξ για όλες τις ε, αναφορές Από πλευρά μα θα συνεχίσουμε να κάνουμε αξιολόγηση των κάθε σε κάθε υπόθεση, ξεχωριστά. Ένα τελευταίο τώρα στοιχείο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Jugendamt. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με κάποιες από τις ε, από τα στοιχεία που ανέφερε ο εκπρόσωπος του Jugendamt. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει ευαισθητοποίηση για τη λειτουργία του Jugendamt, προκειμένου να αποφευχθούν και στο μέλλον υποθέσεις όπου θα υπάρξει ενδεχόμενη παρανόηση, σύγχυση, το... μέχρι ότου ολοκληρωθεί και η αναθεώρηση του Βρυξέλλες 2, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει τεράστια δουλειά, να συνεχίζεται να γίνεται τεράστια δουλειά και να συζητιέται με τα κράτη-μέλη, με τις αρχές, με τους δικαστές, το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η αρχή του συμφέροντος του παιδιού. Και αυτό στη συνέχεια να εφαρμοστεί και στις διαδικασίες που θα αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά το Βρυξέλλες 2 και και θέματα σε επίδοση των αποφάσεων. Σας ευχαριστώ. Να πω δύο λόγια για την ε, αναφορά της κυρίας Μπασφελιέ. Δεν αφορά μέσα το θέμα του Jugendamt, όπως συζητήθηκε και από τους συναδέλφους, αλλά και από τους άλλους αναφέροντες, έχει να κάνει με την ενδεχόμενη αλλαγή του ονόματος. Να πούμε ότι αυτό δεν έχει ακόμα εκδικαστεί ως υπόθεση και πρέπει να το αποφασίσει το δικαστήριο. Είναι δύσκολο λοιπόν. Όταν δεν έχουν ε, πραγματοποιηθεί οι φόβοι ε, αναφέρουσας. Αν όντω συμβεί αυτό που φοβάται η αναφέρουσα, δηλαδή το δικαστήριο το γερμανικό, αποφασίσει ότι η κόρη της θα πρέπει να αλλάξει το επίθετο της από το επίθετο του, της μητέρας στο επίθετο της μητέρας που έχει δεν πρόκειται για το όνομα του πατέρα. Διευκρινίζει εκτός μικροφώνου δυστυχώς η αναφέρουσα. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Δεν το ίδιο είναι το ίδιο, είναι εντελώ διαφορετικό, γιατί δεν θα πάρει του πατέρα το όνομα, θα πάρει το όνομα της νέας συζύγου. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Ναι, ο πατέρας ε, θα ήθελε να αλλάξει το όνομα της κόρης, γιατί και ο ίδιος έχει αλλάξει το επίθετό του, έχει πάρει το όνομα της νέας συζύγου και θέλει να το πάρει και το παιδί. Αυτό, εάν συμβεί, και θεωρεί η αναφέρουσα ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά της, τότε θα πρέπει να κάνετε έφεση σε εθνικό επίπεδο γιατί όπως εξηγήσατε στην αναφορά σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε σχέση με την αλλαγή ονόματος. Αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Ένωση θα μπορούσε να παρέμβει μόνο στην περίπτωση που αλλαγή επωνύμου μπορεί να αποτελέσει πρόσκληση ακόμα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσατε να ασκήσετε έφεση και να αναφερθείτε σε διεθνές συμφωνίες όπως η Σύμβαση της Νέας Υόρκης ή η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εάν υπάρχει τέτοια παραβίαση και θα ζητήσετε, θα μπορούσατε να ζητήσετε από, το Γερμανικό Δικαστήριο να υποβάλει προδικαστικό αίτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα και με παρεμφερή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κατά πόσο μπορείτε να θεωρήσετε ότι πλήτετε το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας του παιδιού σας γιατί ίσως ε, στη Γαλλία η αλλαγή επωνύμου να μην αναγνωριστεί. Δηλαδή αν αλλάξει από, το όνομα από Μπασελιέ σε Γιούργενς δεν αναγνωρίζει ή δημιουργήσει δυσκολίες ε, στις γαλλικές αρχές. Σε αυτή την περίπτωση πλήττεται το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας της κόρης σας όταν θα πρέπει να μετακινηθεί μεταξύ δύο διαφορετικών κρατών μελών. Δεν λέω ότι ισχύει, θα μπορούσατε να επικαλεστείτε τις αρχές και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και μη διάκρισης με βάση την υπηκότητα. Εάν λοιπόν ο Γερμανός δικαστής αποφασίσει ότι πρέπει να αλλάξει το επώνυμο της κόρης σας με το επώνυμο του πρώην συζύγου σας που έχει λάβει το επώνυμο της νυν συζύγου, τότε μπορείτε να επικαλυστείτε και το θέμα του κατά πόσο το δέχεται η κόρη σας. Σε πάση περιπτώσει θα πρέπει να ε, κάνετε προσφυγή σε εθνικό επίπεδο και θα μπορούσατε να ζητήσετε και προδικαστικό ερώτημα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Καλώς, ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα δώσω το λόγο σε τρία μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μου το ζήτησαν. Ένα λεπτό ο καθένας. Οι αναφέροντες επίσης για να κλείσει και το θέμα, γιατί έχουμε 15 λεπτά μόνο. Ο Ενρίκε, ένα λεπτό. Θα είμαι πολύ απαιτητική, δεν θα σας αφήσω παραπάνω χρόνο. Είναι καλό που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, γιατί η κατάσταση στη Γερμανία είναι πραγματικά νομικός πώς πάρα πολύ δύσκολη και ούτε ε, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή ούτε από το παιδί ούτε από τους γονιούς. Εγώ έχω ενημερωθεί και πολλές περιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ε, αυτερεσία των Jugendamt. Εδώ μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος είναι πέρα από το δίκαιο για την εξαγωγή των παιδιών ε, στο εξωτερικό. Πολύ Γερμανοί γονείς και Γερμανοί γονείς ζουν σε μια μεγάλη κατάσταση εξάρτησης και το Jugendamt συχνά πλήττει τους ε, πατέρες συχνά σε ό,τι αφορά την ε, διατροφή. Φυσικά το παιδί αποτελεί παραγόντα ένδυας και είναι δύσκολο το θέμα της καθορισμού του, της διατροφής. Και φυσικά προστίθεται και το θέμα της γλώσσας. Ο κύριος Βίλιαμ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Καταρχάς, να παρακαλέσω να τοποθετηθεί ο εκπρόσωπος του Jugendamt. Τι γίνεται με την ε, μετάφραση και την ερμηνεία σε περίπτωση γονέων που δεν μιλούν γερμανικά. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να πω το εξή. Δεν ε, ξεκαθαρίσαμε ποιες ε, είναι οι παραδεκτές αναφορές, γιατί δεν είμαστε κάποιο υπερδικαστήριο. Το θέμα είναι ότι κάθε εθνικό δικαστήριο συστηματικά κατηγορούν κάποιες αναφορές ότι υπάρχει συστηματική διακριτική μεταχείριση κατά ε, κάποιων συγκεκριμένων ε, επικών. Είμαι ειδικό σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν περιπτώσεις ε, λανθασμένων δικαστικών αποφάσεων. Υπάρχουν λυπηρά στοιχεία και είναι δύσκολα αυτό το θέμα του ποινικού ε, δικαίου σε ό,τι αφορά θέματα ιατρικού ε, δικαίου. Είναι πάντα δύσκολο και φυσικά στα θέματα οικογενειακού δικαίου να δοθούν αποζημιώσει. και παράλληλα αυτά πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η κυρία Σιμπισέσκη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Για λόγους τυπικούς να σας πω ότι ένα τμήμα δικαστηρίου που μόνο ενάντια στους αναφέροντες. Δηλαδή ε, δεν άκουσαν και τα δύο μέρη. Αυτό είναι εντελώ αντιθεσμικό. Εδώ ακούμε μόνο τη μία πλευρά. Και μόνο το, η μία πλευρά θα ακούσει, θα διαδώσει την άποψή της στην κοινή γνώμη. Νομίζω ότι είναι μερολεπτική η διαδικασία. Επόμενη ομιλήτρια. Έχω ένα ερώτημα για τον εκπρόσωπο του Jugendamt, της υπηρεσίας πρόνοιας. Είπατε ότι το, το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να ακούσει τη θέση της υπηρεσίας πρόνοιας. Έχετε όμως στατιστικά στοιχεία σε πόσες περιπτώσεις η απόφαση του δικαστηριού συνάδει με τη θέση της υπηρεσίας πρόνοιας και σε πόσες περιπτώσεις είναι διαφορετική. Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό να το γνωρίζουμε. Πόσες φορές έχει διαφοροποιηθεί το δικαστήριο από τη θέση του Jugendamt. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ και δικαίως και ότι συνήθως ε, όταν τσακώνονται οι γονείς δεν είναι εφικτό να βρεθεί μια αποδεκτή απόφαση από όλους. Θα ήθελα να πω ότι και η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία και η Δανία ε, έχουν και αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν είναι δικαστήριο. Γιατί είμαστε λοιπόν σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρμόδιοι για θέματα ανταλλαγή πληροφοριών, μετεκπαίδευση, σωστά τα είπατε όλα αυτά, ευαισθητοποίηση, όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα κοιτάμε για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και να μην ε, ξυπνάμε, να μην ε, δίνουμε λαθασμένες εντυπώσεις και ελπίδες. Ο κύριος Μάρτιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε ότι είχαν κλείσει αναφορές. Ναι, αλλά θέλω να σα απαντήσω ότι επειδή κλείνει μια αναφορά, αυτό δεν σημαίνει ότι λύνεται και το πρόβλημα. Μπορεί τεχνικά να έχει κλείσει, πολιτικά το πρόβλημα παραμένει. Δεν έχουμε σκοπό εδώ να δικάσουμε μια συγκεκριμένη χώρα αν αύριο υποβληθούν σοριδών αναφορές κατά της Γαλλίας ή της Ισπανίας, με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσουμε. Εμείς είμαστε αποδέκτες χιλιάδων αναφορών για αυτό το ίδρυμα και για αυτή την υπηρεσία πρόνοια στη Γερμανία και παρά την ποιότητα της παρουσίασης σας αγαπητέ εκπρόσωπε δεν απαντήσατε επί της ουσίας. Εμείς έχουμε ερωτηματικά. Απλά μας παρουσίασατε την υπηρεσία πρόνοια στο Γιούγκεντα. Ωραία παρουσίαση κάνατε, σωστά, πράγματι, αλλά δεν απαντήσατε κατά τα λοιπά θα δοθεί συνέχεια. Αν δεν έχετε πρόταση, έχω εγώ πρόταση για το πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά μας. Παρακαλώ. Προτείνω λοιπόν, μετά τη δουλειά στην ομάδα εργασίας, να συμφωνήσουμε πάνω σε μια σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων που θα στείλουμε στις γερμανικές αρχές, εάν συμφωνούν όλοι, και θα ζητούμε συγκεκριμένες ακριβείς απαντήσεις από τις γερμανικές αρχές. Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Και τέλος η Ελεονόρα για ένα λεπτό. Για να δώσουμε το λόγο και στους αναφέροντες. Και εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ότι στην πραγματικότητα δεν έλαβα καμία απάντηση στα ερωτήματα που ετέθηκαν προς τη, τη Jugendamt. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την εργασία, να αποστείλουμε αυτά τα ερωτήματα γραπτός για να ξεκινήσουμε και με μία γραπτή διαδικασία. Πού υπάρχει η έννοια του Ζόργεν Ρέχτ με βάση το οικογενειακό δίκαιο. Δεν έχουμε λάβει ε, απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα όταν μιλάμε για πρόνοια του παιδιού. Αυτό που έχει σημασία είναι να διευρύνουμε το οπτικό μας πεδίο σε σχέση με τα συστημικά στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Φυσικά, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι η βάση της εργασίας μας, αλλά θα πρέπει να διευρύνουμε το πλαίσιο. Ευχαριστώ την Ελεονόρα. Για δύο λεπτά ο εκπρόσωπος του Γιούγκενταμ της υπηρεσίας πρόνοιας και στη συνέχεια δύο λεπτά ο κάθε αναφέρον και θα ολοκληρώσουμε την εξέταση του θέματος. Αλλά δεν ε, μπορούν όλοι οι αναφέροντες, δεν έχουμε χρόνο. Συμφωνήστε για έναν εκπρόσωπο που θα μιλήσει και θα σας εκπροσωπήσει όλους. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο Το θέμα του ονόματο και του επιθέτου. Να σα πω το εξή. Ε, το συζήτησα και με του δικαστέ για τα οικογενειακά ζητήματα και το θέμα λοιπόν θα ήταν ε, να αποφασίσουμε ποια σημασία θα είχε αυτό για το παιδί, όχι για, το, για τη μητέρα. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον ε, το θέμα είναι να καθοριστεί κατά πόσον το παιδί θα ανήκει στη νέα οικογένεια και το θέμα του ονόματος, κατά πόσον ε, θα είχε σημασία. Και τα δύο είναι βάσιμα επιχειρήματα. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως ακόμα και θα πρέπει να το κοιτάξουμε από πλευρά του παιδιού. Το θέμα της ε, γλώσσας. Η γλώσσα εργασίας, η επίσημη στην ε, Γερμανία είναι τα γερμανικά. Το ίδιο ισχύει και στις άλλες χώρες όλα τα πρωτότυπα, όλη η νομοθεσία είναι στα γερμανικά. Όταν στρέφεται κανείς και αποτείνεται στα οικογενειακά δικαστήρια, στο Βερολίνο τουλάχιστον, πρέπει να κάνει τη μετάφραση και το δικαστήριο διαθέτει στο βαθμό του δυνατού ε, μεταφραστές. Διαφορετικές αποφάσεις τώρα μεταξύ Jugendamt και δικαστηρίου δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία γιατί ουσιαστικά το Jugendamt δεν υποβάλλει αποφάσεις προς το δικαστήριο, απλά μια τοποθέτηση δίνει για τις καταστάσεις. Είναι αντικειμενική, ουδέτερη, δεν αποτελεί απόφαση, ούτε περιλαμβάνει απόφαση για τις προτεραιότητες που εντοπίζει. Είναι ουσιαστικά μια βοήθεια προς τον δικαστή. Διαφορετικές αποφάσεις ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λαμβάνονται σε περιπτώσεις ε, ανάθεσης της επιμέλειας όταν είναι διαφορετική άποψη, αλλά είναι σπάνιε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά. Εξ ονόματος των αναφερόντων, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Μικρόφωνο. Please. Γεια σας, είμαι ο γιος ε, της κυρίας Ποτοξοβίτ και θα ήθελα να πω μόνο δύο λόγια σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του κυρίου Γόφμαν. Μας είπε ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των γονέων ε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Jugendamt και λαμβάνει την υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Όταν ήρθε η μητέρα μου στη Γερμανία, ξαφνικά ε, είχε δείξει ενδιαφέρον ε, ο πατέρα μου. Με ρώτησε το Jugendamt πού ήθελα να ζήσω και είπα πολλές φορές ότι ήθελα να είμαι με τη μητέρα μου. Και με ανάγκασαν να κάνω δηλώσεις ξανά και ξανά μέχρι να ακούσουν αυτό που ήθελαν. Ε, δεν με νοιάζει, τους είπα τελικά. Γι' αυτό λοιπόν έχω να πω ότι το Jugendamt είχε αποφασίσει από πριν ότι το συμφέρον μου ήταν να μείνω με τον πατέρα μου. Έτσι λοιπόν προκύπτουν αυτές οι περιπτώσεις παρανόησης. Καλώς. Ακούσαμε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν εδώ και προτείνουμε το εξής. Η ομάδα εργασίας θα συγκεντρώσει τις ερωτήσεις και θα τις απευθύνουμε στις γερμανικές αρχές. σύμφωνα με την πρόταση Μάρτινς. Δεν έχουμε αρμοδιότητα, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαχείριση ως Επιτροπή Αναφορών. Συμφωνείτε? Να ευχαριστήσω θερμά τους αναφέροντες και όλους τους συμμετέχοντες στην πρωινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ.